Colleghi, diamo inizio ai lavori. Καλησπέρα σα. Θα ξεκινήσουμε την ακρόαση αυτή τη συνεδρίαση ε, που είναι αφιερωμένη στην Ένωση για την Μεσόγειο μετά από πρωτοβουλία του συναδέλφου Βενσάου Μπρεγιάου που θα ψηφιστεί, ε, θα παρουσιαστεί μάλλον στην Ολομέλεια του Μαΐου ε, λίγο πριν την ε, Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στη Βαρκελόνη στις 7 Ιουνίου για το ίδιο θέμα. Πριν από κάποιο χρόνο είχαμε την έκθεση του κ. Ναπολιτάνου, η διαδικασία της Βαρκελόνης, Ένωση της Μεσογείου. Και σε αυτή τη φάση συνεχίζουμε τον πολιτικό μας προβληματισμό και αποδεικνύουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή του Εξωτερικών Υποθέσεων επιθυμούν να παρακολουθήσουν εκ του σύνοικης τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Ένωσης για την Μεσόγειο. Δεν χρειάζεται να σας θυμίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νότια ε, περιοχή της που βρέχεται από την Μεσόγειο ε, συνδέεται άμεσα με όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο ευημερία και ειρήνης προς όφελος όλων των πολιτών των κρατών που ανήκουν στην Ένωση της Μεσογείου. Υπάρχουν διάφορες προκλήσεις, ε, περίπλοκες και άρα θα πρέπει να έχουμε το πολιτικό στένος και ένα πραγματιστικό πνεύμα για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις αυτές. Για αυτήν την ακρόαση ο κύριος Πεϊγιάν πρότεινε να εστιάσουμε βασικά σε δύο ε, νέες ε, πολύ σημαντικές πτυχές. Πρώτο είναι οι θεσμικές ε, πτυχές και έπειτα το θέμα των προγραμμάτων και της χρηματοδότησής τους. Για τα θεσμικά ζητήματα είχαμε ζητήσει από τον κύριο Μεζεντέ, τον Γενικό Γραμματέα, τον υποψήφιο Γενικό Γραμματέα, που δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι εδώ, αλλά μας διαβεβαίωσε για την διαθεσιμότητά του να παρέμβει στο μέλλον ενώπιον Τη της Επιτροπής Θα ήταν σκόπιμο να λάβουμε υπόψη αυτή τη δυνατότητα για την πρώτη συζήτηση του κειμένου της έκθεσης. Ήρθαμε λοιπόν σε επαφή με την ε, Ισπανική, Γαλλική και Αιγυπτιακή Συμπροεδρία που λόγω μιας επίσημης άτυπης συνεδρίασης για τα θεσμικά ζητήματα που αποφασίστηκε την περασμένη Πέμπτη και που γίνεται στη Βηρητό, την σήμερα μάλιστα, δεν μπόρεσε να στείλει έναν εκπρόσωπο. Για το τμήμα για τα σχέδια, την χρηματοδότηση και τις επενδύσεις έχουμε μαζί μας δύο προσωπικότητες μεγάλου κύρους που δίχως δισταγμό δέχτηκαν την πρόκλησή μας. Τον κύριο Φοντέν Βιβ Κορτάς που είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τον κύριο Ρίτσαρντ Βεβέρ που είναι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της EuroPaid της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους δύο προσκεκλημένους μας για την παρουσία τους και για την ε, ευγένειά τους, αν είναι σήμερα εδώ μαζί μας και τους ζητώ να παρέμβουν με παρεμβάσεις που να μην ξεπερνούν τα 15 λεπτά έκαστη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκλησή σας και ευχαριστώ και τον συγκητή σας που την πρότεινε την εκδήλωση αυτή. Και το λέω ειλικρινά γιατί νομίζω ότι το 2010 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα έχει ακόμα περισσότερη ειδονή από ό,τι πέρυσι για την ανάληψη δράσεων εκτός της Ένωσης εφόσον ο Μισελ Καμντεσούς το ίδιο αυτό κτίριο αυτήν τη στιγμή παρουσιάζει την έκθεση που θα σας υποβάλει όπως και στην Κομισιόν και το Συμβούλιο και θα προτείνει την αύξηση της αλληλεγγύης μεταξύ Ένωσης και υπολείπου κόσμου μέσω της χορήγησης περισσότερων κονδυλίων εκτός Ένωσης. Επομένως το θέμα αυτό της Ένωσης για τη Μεσόγειο είναι από τις προτεραιότητές μας και αν μου το επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να αρχίσω υπενθυμίζοντας έναν αριθμό απλούστατο Κατά τα 7 τελευταία χρόνια το χρηματοδοτικό μέρος της ΕΤΕ απέφερε πάνω, ε, έδωσε πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ πράγμα το οποίο διευκολύνθηκε ιδιαίτερα από αυτό το εργαλείο που συζητήσαμε και αποφασίσαμε πέρυσι και μας κατέστησε τον πρώτο τραπεζίτη της Μεσογείου. Αυτά από το 2009 ως πρώτο έτος αυτών των δραστηριοτήτων και φέτος θα κάνουμε την τελική συνέντευξη τύπου. Σας λέω όμως ήδη από τώρα ότι υπάρχει, έχουμε σπάσει ρεκόρ δραστηριοτήτων 1,6 δισεκατομμύρια χρηματοδοτήσεων για τις εννέα χώρες της Μεσογείου. Πράγμα που δεν είχε ποτέ του προηγούμενο. Τώρα τα δύο θέματα που θίξατε και εσείς θα τα αναφέρω με ανάποδη σειρά. Πρώτον, πώς μπορεί να συμβάλλει η ΕΤΕ χρηματοδοτώντας την οικονομική ανάπτυξη της Μεσογείου και έπειτα ως απλός τραπεζίτης πώς μπορεί θεσμικά να συμβάλλει όπως σας λέμε τα είπα ανάποδα λοιπόν. αλλά επίτηδες όμως επίτηδες. Λοιπόν, εμείς ε, υποστηρίζουμε τις προτεραιότητες ανατομέα, τις τομεακές προτεραιότητες της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Πέρυσι, όπως σας είπα, δανείσαμε 1,6 δισεκατομμύρια και ε, μέσα σε αυτά, από αυτά το 80% αποτελούν τμήμα των προτεραιοτήτων της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Πρόκειται για κάτι το καινούριο, ένα το πρόσφατο, αλλά ήδη βλέπετε ότι ανταποκρινόμαστε κατά 80% σε αυτά που ζητήσατε μεταξύ άλλων και εσείς και οι υπουργοί που μας αποδώσατε ρόλο συγχρηματοδότη με υπόλοιπους στόχους την απομόλυνση της Μεσογείου σε συνεργασία με την Κομισιόν συντονίζουμε τις δραστηριότητες απομολύνσεως. Οι Υπουργοί ζήτησαν ιδιαίτερα να στηρίξουμε τα θέματα ηλιακής ενέργειας στη Μεσόγειο και τέλος πάλι μαζί με την Κομισιόν το θέμα των θαλασσίων και οδικών λεωφόρων μετακίνησης στη Μεσόγειο. Αυτές οι τρεις προτεραιότητες ε, δεν είναι οι μόνες γιατί προσπαθούμε επίσης να αναπτύξουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουμε για να τα διαθέσουμε στην περιοχή αυτή και τις εγγυήσεις και τα δάνεια αλλά και τη συμμετοχή στο κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων έτσι ώστε να καταστούμε τελικά μέσω των ε, επενδυτικών αυτών ταμείων από τους πρώτους κυριότερους παράγοντες ανάπτυξης στη Μεσόγειο. Γενικότερα δεν προσπαθούμε να βοηθήσουμε να, στην ανάπτυξη της Ιταλο-Ισπανικής πρωτοβουλίας υπέρ των μεσαίων επιχειρήσεων και από τα μέσα Απριλίου ήδη θα σας υποβληθεί η πρώτη μελέτη για επενδύσεις σε χώρες του νότου της Μεσογείου. Ήδη ακόμα συζητάμε με τις χώρες του Μασράκ για να δούμε αν υπάρξει συμφωνία και από τα μέσα Απριλίου θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί τα αποτελέσματα να είναι εκπληκτικά για ορισμένους, ιδίως όσους δεν γνωρίζουν πολύ καλά τη Μεσόγειο. Παραδείγματος χάρη. Είχα την ευχαρίστηση στις 23 Δεκεμβρίου προπαραμονή των Χριστουγέννων στη Ραμαλά να ανακοινώσω τη δημιουργία ενός ταμείου επενδύσεων στην Παλαιστίνη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν την περιφέρεια και που δεν είναι και πολύ γνωστές στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή η επιλογή γιατί επρόκειτο για νέες τεχνολογίες αναπτύσσεται και μέσω της οργάνωσης διασκέψεων όπως την 7η που θα γίνει στην Τίνιδα σε μερικούς μήνες για να αναπτυχθεί και στη Μεσόγειο η ανταγωνιστικότητα. Βεβαίως όλα αυτά τα κάνουμε μέσω, με αρκετά περιορισμένα μέσα και ένα από τα θέματα που τίθεται είναι για σας πώς θα μπορούσαμε να ενδυναμώσουμε αυτή τη στήριξη της Ένωσης προς την Μεσόγειο. Και περνάω έτσι στο θεσμικό τμήμα της παρουσίασής μου. Το Ευρωμεσογειακό Εργαλείο Εταιρικού Διαλόγου και Σχέσης είχε προβλέψει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν να γίνει μέσω της σύναψης εταιρικών σχέσεων μέσα στα υπάρχοντα θεσμικά πλαίσια. Δηλαδή, εμείς έχουμε συμβουλευτικό ρόλο ώστε να φροντίζουμε να χρησιμοποιηθεί η ΕΤΕ ως αναπτυξιακή τράπεζα για τη Μεσόγειο οργανών με διασκέψεις όπως αυτή που ανέφερα για την Τίνιδα που θα γίνει σε λίγο ε, συνεννοούνται μεταξύ τους οι εκπρόσωποι των χωρών μαζί με μας σε ένα κοινό διοικητικό συμβούλιο τρεις-τέσσερις φορές το χρόνο στο Λουξεμβούργο και οι Υπουργοί Οικονομικών συνεργάζονται επίσης όπως θα έκαναν και σε μια ενεργειακή τράπεζα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 18 Μαΐου θα γίνει η επόμενη τέτοια συνεδρίαση εδώ στα Βρυξέλλας. Η εταιρική αυτή σχέση γίνεται λοιπόν με τις ε, χώρες της Μεσογείου αλλά και με τους εκπροσώπους άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που λειτουργούν εκεί. Πρόσφατο παράδειγμα τα εγγένεια τον Οκτώβριο στη Μασαλία μιας καινοτομίας δηλαδή η, Διεθνής, η Παγκόσμια Τράπεζα, η ΕΤΕ και έξι χώρες, εξών πέντε μεσογειακές, η έκτη ήταν η Γαλλία, από κοινού θέλουν να εξυγχρονίσουν τις δημόσιες τους, τον δημόσιο τους τομέα όπως τις μεταφορές και τη συγκοινωνία. Επίσης ελπίζουμε μετά από την έκθεση Καμδεσού που σας υποβάλλεται όπως είπα αυτή τη στιγμή ε, ελπίζουμε να μας ζητήσετε να πάμε ακόμη παραπέρα και να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία αυτή. Ο Ρίχαρδος Βέμπερ νομίζω θα μας το ξαναπεί και αυτός εκ μέρους της Κομισιόν γιατί θέλουμε όσο στενότερη συνεργασία γίνεται με την Κομισιόν για να μην χάνεται χρόνος και βαρύνουν οι διαδικασίες έτσι ώστε το 2010 ό,τι προτάσεις κάνετε να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη στην έκθεση που ευσεβάστως θα υποβάλουμε στο μέλλον. Τέλος, δεν θα ήθελα να καταλήξω εδώ χωρίς να σας πληροφορήσω ότι υπάρχει και μια πρωτοβουλία του Νικολάου Σαρκοζή βάσει της οποίας δημιουργήθηκε μια επιτροπή στην οποία συμμετέχω και εγώ μου ζητήθηκε προσωπικά ανάλυσης μαζί με τον Κάρολο Μιγιό της ιδέας της δημιουργίας μιας πιθανής μεσογειακής τραπέζης για να χρηματοδοτούνται έτσι οι δραστηριότητες της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Πρώτη φορά θα συνεδριάσουν για την ιδέα αυτή στις 8 Μαρτίου, η Εθνή ημέρα της γυναίκας. Και ε, θα γίνει και μια διάσκεψη στις 7 Ιουνίου, όπως ξέρετε, για να καταλήξουμε εκεί όπως ελπίζουμε σε μια τουλάχιστον ενδιάμεση έκθεση τουλάχιστον. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βέμπερ, έχετε το λόγο. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, κύριε και κύριοι βουλευτέ. Κυρίε και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχά να σα ευχαριστήσω ειλικρινά για την πρόσκληση. Είμαστε τόσο ενδιαφέρουσα, αλλά ε, όσο και στρατηγική συζήτηση τη στιγμή που ελπίζουμε ε, να συσταθεί και να αρχίσει να λειτουργεί η γραμματεία προσεχώς τη Ένωση για τη Μεσόγειο. Συνεχίζω από το προαρίσαντα, θα αρχίσω από τα θεσμικά και θα έρθω στη χρηματοδότηση. Για τα θεσμικά. Αλλά εγώ θα ασχοληθώ περισσότερο με τα οικονομικά. Συχνά ακούμε να λέγεται και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε και να διασκεδάσουμε είναι ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο ε, ε, είναι περίπλοκη, δεν είναι πάρα πολύ συνοχή, ε, συνεκτική, είναι συνάρτητη, όχι. όλα αυτά αλληλοσυμπληρώνονται, έχουν μια λογική συνέχεια. Αρχίσαμε από τη διαδικασία της Βαρκελόνης, Βεβαίω προηγουμένω υπήρχαν τα ευρωμεσογειακά πρωτόκολλα. Από εκεί αρχίζει αυτή η προσπάθεια το 1995 με τις τρει πτυχέ τη εταιρική σχέση. Ακολούθησε αυτή η ιδέα, περισσότερο αναπτύχθηκε 2005 με το πενταετέ πρόγραμμα πάντα στα πλαίσια της διαδικασία τη Βαρκελόνη. Στη συνέχεια έχουμε την πολιτική γειτονία που τελικά ήταν μια προσπάθεια εμβάθυνσης και αναζήτηση προ την κατεύθυνση αυτή μετά τη Βαρκελόνη, χρησιμοποιώντα το κεκτημένο τη Βαρκελόνη και εμπλουτίζοντα το. Και τον Αύγουστο έχουμε και μια ε, εκτός από την περιφερειακή προσέγγιση, μια προσέγγιση ένα κράτος και κάθε κράτος επιλέγει ε, να έρθει πιο κοντά στην Ένωση σε κάποιο τομέα ε, περισσότερο ή λιγότερο. Και καταλήγουμε στην Ένωση για τη Μεσόγειο. Και τι είναι η Ένωση για την Μεσόγειο είναι ε, όπως οι ρώσικες κούκλες που μπαίνουν η μία μέσα στην άλλη. Τώρα δεν ε, εφευρίσκουμε τον τροχό από την αρχή, αλλά αναπτύσσουμε και εμβαθύνουμε τις σχέσεις των ε, ευρωπαϊκών χωρών με τις χώρες της Μεσογείου. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ορίσουμε είναι η γεωγραφική περίμετρος. Μιλάμε για 44 χώρες, ενώ 37 είναι χώρες στη γειτονία. Γιατί έχει σημασία αυτό. Γιατί αν κοιτάξουμε μέσω στη χρηματοδότηση που μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή για την Ένωση ή τη Μεσόγειο, διαπιστώνουμε ότι βεβαίως ε, θα πρέπει να καταφύγουμε και στο μέσο γειτονία, αλλά και στο προενταξιακό μέσο, γιατί είναι χώρες στην Ένωση για τη Μεσόγειο που είναι και υποψήφιες χώρες και εντάσσονται στην προενταξιακή χρηματοδότηση. Είτε είναι οι χώρε αυτές οι χώρε πρώην Ιουγκοσλαβία, είτε είναι η Τουρκία. Μπορεί κανείς να το προχωρήσει ακόμα παραπέρα αυτό. Υπάρχουν χώρες στην Ένωση για τη Μεσόγειο που ε, χρηματοδοτούνται σχεδόν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Μέχρι τη Μαυριτανία φτάνει η Ένωση για τη Μεσόγειο. Ε, γιατί ε, η χρηματοδότηση λοιπόν μπορεί να προέρθει από διάφορα μέσα και από την ευρωπαϊκή σκοπιά είναι πολύ ευρύτερη ε, από ό,τι κανείς θα θεωρούσε. Δεν είναι μόνο το μέσο γειτονία. Τα ίδια ισχύουν και για το πολιτικό, νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Πάντα όμως για τη χρηματοδότηση. Ε, και πάλι έχουμε αλληλοσυμπλήρωση όλων των ε, προσπαθειών, διότι τα έργα που χρηματοδοτούνται ως προτεραιότητα εντάσσονται και στην πολιτική γειτονία προ τον Νότο ή στην ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση. Δεν έχουμε, όχι μόνο δεν έχουμε ασύμβατο ούτε επικαλύψει, το αντίθετο, εμβάθυνση και ανάπτυξη και επέκταση όλων αυτών των προσπαθειών. Είναι σαφές ότι ε, στα χρηματοδοτικά το, η βάση που έχουμε είναι ε, το μέσο γειτονίας. Ο κύριος ε, μίλησε για τα σημαντικά δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μελλοντικά και ισχύοντα. Ε, εμείς ξέρετε ότι έχουμε για μια επταετή περίοδο 12 δισεκατομμύρια και από τα 12 δις περίπου τα 2 τρίτα, 10, αφορούν τις χώρες της Μεσογείου. Και θα ήθελα να θυμίσω εδώ, ε, κατά συνέπεια, ε, συνεχίζοντας από τα όσα είπα προηγουμένως, ότι οι χώρες αυτές που θα συμμετέχουν ε, θα χρηματοδοτούν εν μέρη την προσπάθεια αυτή. Είπαμε ότι υπάρχουν χώρες που είναι υποψήφιες και μπαίνουν στην προεταξιακή διαδικασία και έχουν ένα ποσό αντίστοιχο στην μεγέθους με την πολιτική γειτονία και μπορούν και από εκεί να αντιληθούν κονδύλια για κάποια έργα της Ένωσης ή τη Μεσόγειο. Γιατί έχει σημασία αυτό. Γιατί. Σε αντίθεση με κάποιες ιδέες που ακούμε δεξιά και αριστερά, για τη μεσογειο γιατι εχει σημασια αυτο σε αντιθεση με από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για την Ένωση για τη Μεσόγειο είναι η ίδια περίπου με την πολιτική γειτονία. Ακόμα και αν η οικοδόμηση γίνεται με βάση κάποια έργα συγκεκριμένα. όπως ιστορικά έγινε για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, χρήματα υπάρχουν, αρκούν, ε, όχι βέβαια, προφανώς και δεν αρκούν. Ε, οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστιες. Η δυνατότητα απορρόφησης των χωρών αυτών της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου συχνά χαρακτηρίζεται ανεπαρκής η απορροφητικότητα η λεγόμενη. Δεν χρειάζεται να είναι κανεί πολύ παρατηρητικός για να διαπιστώσει ότι είναι τεράστιε οι ανάγκε υποδομών, τεράστιες, κατάφορε, κραυγαλές. Ε, είναι δεδομένες οι ανάγκε και στο περιβάλλον και στην απορρίπανση τη Μεσογείου και στην ενέργεια. Υπάρχουν οι ανάγκες, είναι γνωστές. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να βρούμε και τα χρήματα πώς τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα εστιαστούν στις προτεραιότητες και να γίνουν κοινέ προσπάθειες με συγχρηματοδότηση και από άλλους πόρους. Θα πρέπει να βρούμε τώρα εκείνη την, την οικονομική κατασκευή, ας πούμε, και αυτό θα κάνει η γραμματεία και ελπίζουμε σε λίγες εβδομάδες ή μήνες στη Βαρκελόνη να γεννηθεί αυτή η γραμματεία. Λοιπόν, εκεί θα ε, δράει η γραμματεία αυτή ως πύργος ελέγχου τρόπο για την Ένωση για τη Μεσόγειο και τα όσα θέλουμε να κάνουμε. Καλά λοιπόν τα θεσμικά, αλλά τα συγκεκριμένα είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί η ιδέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο είναι συγκεκριμένα ε, σχέδια και έργα να κάνουμε. Με την ε, Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και με διμερή συνεργασία και μιλώ για, δάν, για ε, δωρεέ εδώ όχι δάνεια, και από την ιδιωτική πρωτοβουλία μπορούμε να κινητοποιήσουμε με σύμπραξη ε, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τις λεγόμενες ΣΔΙΤ, για τα έργα υποδομής, για τις επενδύσεις που είναι τεράστιες και θα πρέπει να κινητοποιηθεί και ο ιδιωτικός τομέας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση ισχυρή, δημόσια δέσμευση ισχυρή και βεβαίως να ε, έχουμε ε, ε, τέτοιες οικονομικές κατασκευές ώστε να είναι ε, τα έργα και βιώσιμα αλλά και να μπορούμε να τα πουλήσουμε, να τα προβάλλουμε στον ιδιωτικό τομέα, να τα υποστηρίξει. Έξω και οι τράπεζε επενδύσεων, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, υπάρχουν και διμερείς συνεργασίες όπως είπαμε, όπως είναι στη Γερμανία, η ΚΑΕΦΒ, η ΑΕΦΔ στη Γαλλία και η υπηρεσία για την αναπτυξιακή συνεργασία που έχει η Ισπανία κτλ. Υπάρχουν λοιπόν ε, τέτοια χρηματοδοτικά ιδρύματα ε, που μπορούν να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή. Πώς θα έρθει λοιπόν η λύση σε αυτά τα προβλήματα, σε αυτά τα σχέδια και πώς θα είναι επιτυχής η λύση αυτή. Ο πρώτο στάδιο, σας είπα, είναι να στηθεί πολύ γρήγορα η γραμματεία, να στελεχωθεί ε, παρκώς και από πραγματογνωμοσύνη και από ανθρώπινο δυναμικό, να υπάρχει πολιτική όθηση και βούληση από τη στιγμή που θα συσταθεί η γραμματεία έτσι ώστε να προχωρήσει η δουλειά ταυτοποίησης, ε, εντοπισμού που έχει ήδη αρχίσει και να αρχίζει να τρέχει η χρηματοδότηση, τουλάχιστον στο χαρτί, και να κινητοποιηθούν οι διάφοροι φορείς, είτε είναι ε, το δημόσιο, ε, ευρωπαϊκά χρήματα, ιδιώτες ε, και οι τράπεζες και τα κράτη-μέλη. Υπό τις συνθήκες αυτές μπορεί κανείς να φανταστεί ότι θα ευδοκιμήσει πολύ γρήγορα η Ένωση για τη Μεσόγειο. Είχαμε κάποιες αρχικές τριβές και καθυστερήσεις στην πυροδότηση, αλλά δεν σημαίνει ότι θα συνεχιστεί αυτό. Έχουμε προβλήματα, τα βλέπουμε όλοι, καμιά φορά οδηγεί αυτό σε καθυστερήσεις, ε, μέχρι και σε ακυρώσεις συνεδριάσεων, αλλά θα έρθω να διαπιστώσω το εξής, διότι εμείς ασχολούμαστε με την πολιτική γειτονίας. Στην Ανατολή έχουμε αρχίσει τη συνεργασία και λειτουργεί καλά και μάλιστα ξεκίνησε μετά την Ένωση για τη Μεσόγειο. Είναι λοιπόν καιρός να κοιτάξουν όλες οι ενεχόμενες χώρες τι συμβαίνει προς Ανατολάς. Εμείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε υπέρ μιας ισόρροπης πολιτικής γειτονίας και είναι εξίσου σημαντική Ανατολή με τον Νότο και Τούμπαλιν, αλλά προς το παρόν αφήνουμε να διαπιστώσουμε ότι προχωράει η διαδικασία πιο γρήγορα ανατολικά. Ε, και ποιο μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι μικρότερα τα προβλήματα στην Ανατολή. Είχαμε το πρόβλημα στη Γεωργία και ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν στον Κάφκασο και λίγο παραπέρα. Ε, και αυτά δεν είναι κρίσιμα και καμιά φορά πιο δύσκολα από άλλα της Μεσογείου. Τελειώνω με την ερώτηση αυτή και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βέμπερε. Ο πρώτος που παίρνει το λόγο είναι ο εισηγητής ο κύριος Πεγιό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Φοντενοβίβη και τον κύριο Βέμπερ για την ε, παρουσία τους εδώ που δέχτηκαν δηλαδή την πρόσκλησή μας και σας ευχαριστώ για την ε, προσήλωσή σας ε, στη δράση αυτή αλλά αυτό φαίνεται και από τα όσα είπατε. η στάση και η θέση του Ευρωκοινοβουλίου και εδώ και αναφέρομαι στο συμπέρασμά σας κύριε Βέμπερ είναι να επιμείνουμε στην ανάγκη στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποίησης που ε, οικοδομείται γύρω από διάφορα σύνολα χωρών, να φτιάξουμε μέσα σε αυτού του προγράμματος του Μεσογειακού ένα χώρο ειρήνης και ευημερία για το μέλλον. Βέβαια και την απουσία ε, θεσμικών ε, εκπροσώπων ε, που ενδιαφέρονται άμεσα για το θέμα και ελπίζω πως θα μπορέσουμε σύντομα να το καλύψουμε αυτό το κενό μας είπαν σύντομα πως ε, η κοίηση της ε, ιδέας αυτής για την Ένωση για τη Μεσόγειο δεν ήταν εύκολη αλλά ελπίζουμε πως τουλάχιστον το Μάρτιο όλα αυτά θα τοποθετηθούν σε γερές ε, στέρεες βάσεις. Εν πάση περιπτώσει, στην προετοιμασία τη διάσκεψη κορυφή του Ιουνίου, το Ευρωκοινοβούλιο θέλει να δώσει κάποιε κατευθύνσει και ταυτόχρονα να δείξει πω υποστηρίζει στεναρά τόσο το θεσμικό εγχείρημα όσο και το πολιτικό. Και ε, πίσω από όλα αυτά την ανάγκη να βρεθεί, γιατί είναι το μέγα ζήτημα που τίθεται, να βρει την απαραίτητη χρηματοδότηση και τα συγκεκριμένα προγράμματα, τα κατάλληλα προγράμματα. Έχω κάποιες ερωτήσεις, ε, κύριε Φούντεβίβ, να σα θέσω άμεσα. Είπατε πως ε, ήσασταν ο πρώτο επενδυτή στην Μεσογειακή ζώνη. Μπορείτε να μας δώσετε μια κατάσταση προόδου όσον αφορά τους άλλους επενδυτές. Δηλαδή, σήμερα επειδή ίσως να υπάρχει μια σχετική μείωση των ευρωπαϊκών επενδύσεων, ποια είναι η παρουσία των Αμερικανών, των χωρών του Περσικού κόλπου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, το αναφέρατε επίσης, είστε υπεύθυνο για τον συντονισμό των τριών από τα έξι προγράμματα προτεραιότητας και επίσης ε, το αφήσατε να εννοηθεί στην παρέμβασή σας. Μήπως μπορείτε να μας πείτε ποια είναι επίσης η κατάσταση προόδου αυτών των προγραμμάτων, ποια είναι τα χρονοδιαγράμματά τους, η χρηματοδότησή τους και πώς προχωράει αυτή η συντονιστική εργασία. Και τέλος, ε, ίσως μας είπατε πως ε, προσωπικά ασχοληθήκατε, είναι όμως ένα σχέδιο παλιό, ακόμα και αν ο πρόεδρος σας όρισε. Πάντως υπάρχει αυτό το σχέδιο για μια ευρωμεσογειακή τράπεζα. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω, δηλαδή ποια θα ήταν η προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας ευρωμεσογειακής τράπεζας και επίσης να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν διάφορους, από όσο γνωρίζω, να είναι δυσμενοί σε σχέση με αυτήν την πρόταση και κυρίως τους Ευρωπαίους εταίρους που είναι αρνητικοί τέταρτη ερώτηση και ξέρω πως ε, βρίσκεται μέσα στις ανησυχίες πολλών. Μήπως μπορείτε να μας υποδείξετε σε σχέση με τις επενδύσεις ποιοι είναι οι παράγοντες ε, που καθυστερούν ή που εμποδίζουν τη χρηματοδότηση και αν θα είχαμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τα πράγματα γιατί διάφορα προγράμματα έχουν ξεκινήσει για την διασφάλιση των επενδύσεων αλλά θα ήθελα να γνωρίζω την άποψή σας ως τραπεζικού για αυτό το θέμα. Κύριε Βέμπερ, είπατε διάφορα πράγματα, αλλά αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και πίσω από τα όσα είπατε, τα όσα κρύβονται, είναι να ανησυχώ. Γιατί με τις άποψεις, πως, και είναι άποψη και του Κοινοβουλίου, πως δεν υπάρχουν απαραίτητοι πόροι για το πρόγραμμα αυτό. Γνωρίζετε πως η θέση του Ευρωκοινοβουλίου, που ήδη είχε την ευκαιρία να εκφραστεί, είναι πως η οικονομική συμβολή της ε, Ένωσης ε, θα πρέπει να γίνει χωρίς ε, άλλη σχέση, σχέση μάλλον με τις υπόλοιπες επενδύσεις που μπορεί να γίνουν στον χώρο. Εάν τώρα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με τον προϋπολογισμό, σήμερα το είπατε πως είναι ανεπαρκής και πώς προβλέπετε τις δημοσιονομικές προοπτικές για το 2014-2020. Έπειτα, υπάρχει νομίζω επίσης ανησυχία σε σχέση με την Γενική Γραμματεία. Εγώ, σας το είπα κατηδίαν, θεώρησα πως ήταν κακό σύμβολο το να πρέπει να συζητήσουμε σήμερα την ε, του Γενικού Γραμματέα και τον απληρωτή Γενικού Γραμματέα και να ορθολογήσουμε, εξορθολογήσουμε μάλλον τους αμοιβέ της Γενικής Γραμματείας. Αλλά γενικότερα, και θα ήθελα να έχω την άποψή σας ε, εδώ, αν πιστεύετε ότι αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ που είναι ο που κυκλοφορεί για την χρηματοδότηση της λειτουργίας τη Γενικής Γραμματείας αρκεί και τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν. Υπάρχουν ήδη άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης. Και τέλος, γιατί μέσα στην ιστορική αναδρομή που μας κάνατε και εμείς συμμεριζόμαστε την άποψη πως η διαδικασία και η δημιουργία της Ένωσης για την Μεσόγειο είναι μέσα στη συνέχεια των όσων έχουν γίνει παλαιότερα, ποια θα είναι η οργάνωση της εργασίας ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία και την Κομισιόν. Πώς προβλέπετε να λειτουργήσουν τα πράγματα για την ώρα. Ευχαριστώ και τους δύο που θα μας διαφωτίσετε για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε, κύριοι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τέσσερα πολύ μεγάλου εύρους ερωτήματα. Για να απαντήσω πλήρως θα έπρεπε να ξεπεράσουμε κατά πολύ τη συνεδρίαση αυτή. Ρωτήστε ποιοι είναι οι άλλοι επενδυτές στη Μεσόγειο εκτός από την ίδια την Ένωση μαζί με την ΕΤΕ και την Κομισιόν κτλ. Υπενθυμίζω ότι το πρώτο στοιχείο της χρηματοδότησης είναι τα εμβάσματα των μεταναστών και μεταναστριών. Αυτοί οι μετανάστες είναι που έχουν έρθει και εργάζονται στην Ευρώπη που στέλνουν τα εμβάσματά τους στις χώρες της Μεσογείου. Και αυτό είναι δύσκολο να μεταφραστεί σε επένδυση. Δεύτερον, ένα στοιχείο μείωσης των επενδύσεων, τα οι άμεσες επενδύσεις από τρίτους εκτός Ένωσης. Όταν μειώνονται οι επενδύσεις είναι προφανές ότι η ανάπτυξη μειώνεται. Σε ζώνες εκτός Ένωσης λοιπόν, ποια είναι η σχετική σημασία των κεφαλαίων προέλευσης Περσικού κόλπου ή Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Περσικός είναι θέμα που συζητιέται συχνά αλλά συνήθως οι επενδύσεις εκεί γίνονται στα ακίνητα. Λιγότερο καινοτόμες επενδύσεις, δηλαδή λιγότερο παραγωγικές και προσπαθούμε ένα τμήμα των επενδύσεων αυτών μέσω της Ισλαμικής Αναπτυξιακής Τράπεζας να, τα μετακινήσουμε σε... και σε άλλους τομείς, αλλά είναι σχετικά δύσκολο. Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται επίσης για, μέσω των αμέσων ε, ξένων τρίτων επενδύσεων αλλά δεν συμφωνούν όλα αυτά με το στόχο της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άλλο ερώτημα, πώς συντονίζονται οι τρεις στόχοι που μας εμπιστευτήκανε για την απομόλυνση έχει γίνει ο απολογισμός. Έγινε μια μελέτη δηλαδή για το βαθμό μόλυνσης στη Μεσόγειο και τις τοποθεσίες της μεγαλύτερης μόλυνσης και θα δούμε λοιπόν πού και πώς πρέπει να εφαρμοστούν ε, μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος με πρότυπα ευρωπαϊκά. Άρα θα χρειαστεί μεγάλη επένδυση μέχρι το 2020 και άρα χώρα με τη χώρα θα επενδύσουμε στην απομόλυνση των παραλιών. Για τις θαλάσσιες μεταφορές και τις οδικές όμως υπάρχει μία χάρτα, πρόγραμμα προτεραιοτήτων στις επενδύσεις και πρέπει τώρα να την εφαρμόσουμε προοδευτικά τη χάρτα αυτή. Για τις οδικές μεταφορές νομίζω ότι το πιο προχωρημένο σχέδιο θα το δούμε όμως ξανά στις 7 Μαρτίου κατά τη διάσκεψη Μαρόκο Ένωσης είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης του Ισυπερταχίας, Ταγκέρης και Νίτρα και για τα λιμάνια για τα λιμάνια λέγω έχουμε μελετήσει τα πράγματα για να δούμε πώς θα μπορούσαν τα μεσογειακά λιμάνια να συνδεθούν περισσότερο με την ενδοχώρα και μάλιστα με τρόπο που να σέβεται την προστασία του περιβάλλοντος. Μου ζητήσατε επίσης ένα σχόλιο για την Μεσογειακή Τράπεζα. Γιατί δεν υπάρχει ήδη ποια θα ήταν η σημασία της και γιατί κανείς δεν το σκέφτηκε μέχρι τώρα. Η αξία της θα ήταν να επιτρέψει στις μεσογειακές χώρες να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις χώρες της Ευρώπης και να επιτρέψει παραδείγματο χάρη την έκδοση ομολόγων σε τοπικό νόμισμα είναι δηλαδή θέμα δίκαιας εκπροσώπησης των μεσογειακών χωρών κατά κάποιο τρόπο. Γιατί κανείς δεν το σκέφτηκε μέχρι τώρα για δύο κύριους λόγους που δεν έχουν σχέση με λεπτομέρειες. Ο ένας είναι ότι έπρεπε να αποδειχτεί πρώτα ότι η δημιουργία μιας τέτοιας τράπεζας δεν θα αύξανε το κόστος της λειτουργίας των αγορών και ο δεύτερος είναι ότι έπρεπε να βεβαιωθούμε πρώτα ότι θα χρησιμοποιούσε καινούργια κεφάλαια. Όχι απλώς επαναχρησιμοποίηση ήδη υπαρχόντων ταμείων, γιατί τότε δεν έχει καμιά σημασία η ύπαρξη μιας τέτοιας τράπεζας. Αν αντίθετα έχει πρόσθετα δημόσια κεφάλαια ή ιδιωτικά, τότε θα είχε κάποιο νόημα. Τέταρτο ερώτημα, κάποια οικονομική ανάλυση του αποπαγώματος των επενδύσεων. Όλες οι χώρες αυτές, η κάθε μία είναι πολύ μικρή για να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις. Ενώ μόνο όλες μαζί μπορούν να το κάνουν, σε συνεργασία βέβαια με την Ένωση. Φυσικά είναι λιγότερο σαφές για την Αίγυπτο αυτό από ό,τι για τις άλλες χώρες γιατί είναι η μεγαλύτερη εσωτερική αγορά η Αιγυπτιακή αλλά για όλες τις υπόλοιπες χώρες η περιφερειοποίηση της πολιτικής μας είναι κάτι το πρωτεύον για να αποπαγωθούν οι επενδύσεις, οι διεθνείς επενδύσεις. Υπάρχει και ο κίνδυνος των ισοτιμιών. Οι επενδύσεις σε χώρες όπου δεν είναι γνωστό αν οι σχέσεις του τοπικού νομίσματος με το ευρώ δεν θα διακυμανθούν με τρόπο που να μη συμφέρει στον επενδυτή είναι ένας λόγος αποφυγής. Άλλο, καμία από αυτές τις χώρες μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει δημοσιονομικό εξυγχρονισμό ανάλογο με αυτόν που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό σημαίνει ότι συνολικά η αποταμίευση που υπάρχει στις μεσογειακές χώρες δεν μετατρέπεται σε μακροχρόνιες επενδύσεις λόγω ακριβώς του φόβου που υπάρχει να μην είναι αποδοτική διότι μόνον ένας διεθνώς αποδεκτός οικονομικός παράγων θα μπορούσε να το κάνει. Δεν υπάρχουν μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκεί που να επιτρέπουν τη μετατροπή του χρήματος σε επένδυση. Α, πολύ ωραία απαντήσω για την ερώτησή σας αν τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι επαρκή. Τουλάχιστον όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό στο πλαίσιο των κονδυλίων που έχουμε, είμαστε μπλεγμένοι στο μηχανισμό των δημοσιονομικών ε, προοπτικών και του δημοσιονομικού πλαισίου και άρα είναι προφανέ ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτού του κανόνε. Ο διαθέσιμος, η διαθέσιμη όγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε είναι για την ε, είτε είναι για την ε, Μεσόγειο και για τι υπόλοιπε πολιτικέ, ε, ξέρετε ποια είναι τα ποσά. Τώρα για τα κράτη-μέλη και τι διμερείς του επαφέ και για τι αναπτυξιακέ του πιστώσει που είναι αφιερωμένε στη Μεσόγειο ακριβώ την ίδια απάντηση θα σα δώσω. Και εκεί υπάρχουν ε, προγραμματικές προγραμματικά κονδύλια και θα έλεγα πως η χρηματοπιστωτική κρίση έχει επηρεάσει όλες τις χώρες μας και ξέρουμε σε ποιο βαθμό σε επίπεδο δημοσιονομικών ελλημάτων και χρέωσης ε, και χρέους ε, έχουμε προβλήματα, οπότε πολύ δύσκολα δεν είναι καλό το κλίμα για παραπάνω χρηματοδότηση στους επόμενους μήνες και ε, χρόνια. Στο επίπεδο των τραπεζών η ΕΤΕ ε, πολύ σύντομα θα αναθεωρήσει την εξωτερική της αναπτυξιακή βοήθεια και ελπίζουμε όλοι πως θα αυξηθεί, τουλάχιστον από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε πως θα το ακολουθήσουν και τα κρατημέλη αυτή την ευχή. Ε, αλλά βέβαια είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο. Θα πρέπει βέβαια εκεί να προσθεθούν και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπουν οι διμερείς άλλοι φορείς, είτε η Παγκόσμια Τράπεζα, είτε η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, είτε τα άλλα διμερεί όργανα όπως η ΚΑΕΒ, e η ΕΦΔΕ, η ευσύ της του Ισπανικού Οργανισμού και ούτω καθεξής, γιατί είναι πολύ σημαντικό όλοι να προσπαθήσουν να συνεργαστούν. Και έχουμε επιτυχία σε αυτό το επίπεδο με την ΕΤΕ, οι συνάδελφοι των άλλων τραπεζών, των πολυμερών και εθνικών τραπεζών, ε, είτε μέσω εργαλείων όπως η διευκόλυνση γυπνίασης που φτιάξαμε πριν από 18 μήνες και με την ΑΕΦΤΕ, την ε, ΚΑΕΦΒ και την ΡΕΤΕ μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε με πάνω από 5 δις επενδύσεων σε 18 μήνες, ε, συνδυάζοντας και συνδιοργανώνοντας όλες μας τις προσπάθειες ε, και μοιράζοντας και τα έξοδα. Τις δαπάνες. Αυτό είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Βέβαια, αυτή τη στιγμή τα κονδύλια είναι περιορισμένα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και απέναντί μας έχουμε τεράστιες ανάγκες. Και γι' αυτό και θα πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να κινητοποιηθεί ο ιδιωτικό τομέα. Και ο κύριος ε, Φοντέν Βίβ το είπε ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει φιλοσοφία ε, ε, Ευεργέτη θέλουν να κάνουν επενδύσεις, ε, να είναι εξασφαλισμένες αυτές οι επενδύσεις και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν ε, αγορές αρκετά ευρείες. Δεν φτάνει μια μικρή αγορά 10 εκατομμυρίων για να δικαιολογήσει μια σημαντική επένδυση. Θα πρέπει επίσης να εγγυηθούμε την νομική ασφάλεια αυτών των επενδύσεων με μια εμπορική διακυβέρνηση και νομική που να είναι κατάλληλη, που να προστατεύει φυσικά τις επενδύσεις που γίνονται σε νομικό ε, και χρηματοπιστωτικό επίπεδο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι ε, παραπληρωματικά και θα πρέπει να συνδυάζονται. Όσον αφορά την οικονομική συμμετοχή της Ένωσης, τι θα κάνουμε στο μέλλον ε, για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020. Αυτή είναι η συζήτηση που έχει ήδη ξεκινήσει και που θα γίνει όλο ένα και πιο καυτή τους επόμενους μήνες και έτη και εδώ θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση και γνωρίζουμε πως η κατάσταση δεν είναι πολύ ανθυρή. Αλλά αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Αν τα κρατημέλη το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θεωρήσουν πως η γετνίωση είναι ε, κάτι που αξίζει να έχει την προτεραιότητα και να έχει ιδιαίτερη προσοχή, τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να το αποφασίσουν και ως ε, δημοσιονομική αρχή έχετε πολύ σημαντικό ρόλο να παίξετε ώστε αυτές οι προτεραιότητες να μετατραπούν σε ποσά, σε κονδύλια. Για τη Γενική Γραμματεία, 10 εκατομμύρια ευρώ αρκούν. Όλα εξαρτώνται από το τι θα κάνει ο Γενικός Γραμματέας και ποια θα είναι η περίμετρος δράσης του. Το θέμα της δημιουργίας ενός νέου θεσμού είναι ότι κάθε φορά είναι το πρόβλημα του προσωπικού, το νομικό, της θέσπισης, της λειτουργίας και ούτω καθεξής. Θα ήταν κάπως κοινικό να το πω εγώ από μέρο μου ότι όταν δεν έχουμε πολύ χρόνο δημιουργούμε μια δομή. Σημαίνει ναι. ότι μπορούμε έτσι κάλλιστα να καθυστερήσουμε, να περάσουμε το χρόνο μας, ωστόσο η συγκεκριμένη γραμματεία είναι απαραίτητη και θα πρέπει να γίνει λειτουργική. Για να γίνει λειτουργική λειτουργική θα πρέπει να έχει τον κατάλληλο προπολογισμό, λειτουργικό προπολογισμό και έπειτα ένα μήνυμα με επιχειρησιακού προπολογισμού. Γιατί το να κάνουμε διάφορε χρηματοπιστωτικέ ακροβασίε και να βάζουμε ε, διάφορα προγράμματα προτεραιότητα, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν με εμπειρογνωμοσύνη κανονικά και με έρευνε. Αυτά κοστίζουν πολύ ακριβά. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι ένα κούφιο κέλυφο όλα αυτά που δεν θα κάνει τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν τα επαρκή μέσα. 10 εκατομμύρια ίσως να είναι τσίμα τσίμα στο πλαίσιο των όσων μπορούμε να φανταστούμε. Πώς θα συμβάλλει τώρα η Κομισιόν θα συμβάλλει, γιατί έχει αποφασίσει ότι θα συμβάλλει. Όλα θα εξαρτηθούν από το μέγεθος του προπολογισμού, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε το κονδύλι για το οποίο μιλάμε. Εγώ προσωπικά πιστεύω πως είναι υγιές να διατηρηθεί αυτή η αρχή, ότι να συμβάλλουν όλες, όλα τα μέρη, γιατί πιστεύω πως αν θέλουν να δείξουν την πολιτική σημασία που προσδίδουν στο θέμα, είναι να βάλει ο καθένας ε, το δικό του κομμάτι. Δηλαδή όλοι ξέρουμε πως οι μεσογειακοί εταίροι μας δεν έχουν τα ίδια μέσα όπως έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες και σίγουρα και με ανάμεσα ευρωπαϊκές χώρες ε, υπάρχουν διαφοροποίησεις. Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας να βάλει το χέρι στη τσέπη όσο μπορεί για να αποδείξει πως είναι έτοιμος να κάνει προσπάθειες για να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτή η ένωση. αν θα πρέπει ο καθένα να χρηματοδοτεί του δικού του υπαλλήλου ή του αποσπασμένου του υπαλλήλου στην γραμματεία. Εγώ προσωπικά ω μάνατζερ ε, θα σα πω ότι όσο πιο περίπλοκο είναι το θέμα, τόσο λιγότερο λειτουργεί. Όσο πιο απλό είναι, τόσο καλύτερα. Εγώ θα προτιμούσα να, δίνουν, να παίρνουν όλοι την ίδια αμοιβή για την ίδια εργασία και έπειτα θα προτιμούσα να έχω εγώ τη διαχείριση των πόρων μου. Αυτό είναι μια κοινή λογική, δηλαδή μπορεί ένας να έχει τα πάντα στη διάθεσή του και ο άλλος να μην έχει στη λόγια να γράψει, να ε, μπορούν όλοι να δουλέψουν μέσα στις καλύτερες συνθήκες και να έχουν και μια νομική ασφάλεια. Ε, στο επίπεδο της καθημερινής ζωής. Μια γραμματεία λοιπόν ναι, λειτουργική, επιχειρησιακή, με τα απαραίτητα μέσα που θα τους επιτρέπουν να κάνει τη δουλειά της και την επιχειρησιακή. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Βέμπερ. Α, συγγνώμη, ξέχασα την τελευταία ερώτηση να απαντήσω. Δηλαδή το πώς θα διοργανωθεί, συγγνώμη. Δύο λόγια. Ε, η συνεργασία μεταξύ Κομισιόν και Γραμματείας. Είναι σαφές ότι αν θέλουμε να συνεργαστούμε, η Γραμματεία της Βαρκελόνης, η Κομισιόν Εξορισμού είναι στις και άρα χρειάζονται κάποιες αποσπάσεις. Τουλάχιστον κάποιος από την Κομισιόν να πάει στη Βαρκελόνη. Και θα έλεγα ε, πως ε, θα πρόκειται για μια επιχειρησιακή γραμματεία χρειάζονται τουλάχιστον δύο ειδικοί, ένας πολιτικός και ένας επιχειρησιακός, γιατί να φτιάχνει κανείς ε, προγράμματα δεν είναι το ίδιο με τη διοργάνωση υπουργικών διασκέψεων και η δική μου προσωπική άποψη, προσωπική άποψη επιμένω, γιατί είμαι βέβαιο πω αν βάλουμε την ερώτηση στην Κομισιόν θα πούνε σίγουρα όχι, αποκλείεται δύο άτομα, πάντως κανονικά για να είναι σωστά οργανωμένα θέλουμε δύο ανθρώπους στην Βαρκελόνη. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω τώρα με μια σύντομη δική μου ερώτηση για τις κλιματικές αλλαγές. Ποιες θα, ποιες θα μπορούσαν να είναι οι ε, επιπτώσεις για τη Μεσόγειο. Ήδη φαίνονται κάποιες και τώρα θα δώσω λόγο στον Πιέρ Αντώνιο Παντζέρη. Ε, Πόσο ε, χρόνο έχω στη διάθεσή μου, γιατί 45 λεπτά. Όχι, εγώ θέλω να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Εσείς ε, ε, δείξατε κάποιους ε, δρόμους που ακολουθούμε, ωστόσο πιστεύω πως ένα, σε ένα βαθμό οι προσπάθειες που γίνονται, το πλαίσιο είναι καθοριστική σημασία. Σίγουρα έχουν γίνει πρόοδοι από την άποψη των διμερών σχέσεων, των οικονομικών, ε, διάφορες χώρες ε, στην περιοχή αναπτύχθηκαν οικονομικά πολύ καλύτερα από ό,τι προβλεπόταν, αλλά το πλαίσιο αναφοράς δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό και τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι τώρα συχνά είναι απογοητευτικά. Έχω την εντύπωση πως σε πολλές χώρες από τον ευρωμεσογειακό χώρο έχουν χάσει το τρένο και δυσκολεύονται να, ξανα, να το ξαναπρολάβουν. Εγώ πιστεύω πως ήταν πολύ χρήσιμο να διαπιστωθούν οι δυσκολίες. αρκεί να θυμίσουμε τη διαδικασία της Βαρκελόνης, γιατί τώρα φτάνουμε στη 15 ετία, αλλά οι στόχοι που είχαν εντοπιστεί τότε σε αυτήν τη διαδικασία δεν έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό και δεν διαβλέπουμε να υπάρχουν καν οι προϋποθέσεις για ανάκαμψη. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη του τι, το τι ε, διακυβεύεται σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, υπάρχει το θέμα το σημερινό, αλλά ε, Μέση Ανατολή, ο Λίβανο. Ε, ε, ψυχρός πόλεμο ανάμεσα στην Αλγερία και στο Μαρόκο, που καθυστερούν όλη τη διαδικασία. Όλε αυτέ οι χώρε είναι διαφορετικέ μεταξύ του. Εσεί μιλήσατε για περιφερειοποίηση, αλλά ενώ υπήρξαν πρόοδοι σε κάποιου τομεί, σκέφτομαι α πούμε από το Μερκοσούρ μέχρι την Ασία, εδώ δεν μπορούμε καν να φτιάξουμε ένα περιφερειακό πρόγραμμα συνεργασία. Το πρόβλημα αυτών των χωρών, μάλλον είναι αυτών των χωρών, αλλά αφορά και την Ευρώπη, αν θέλουμε να έχουμε ένα μήνυμο σταθερότητα και οικονομικής ανάπτυξης. Κάτι άλλο πάνω στο οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε εμείς, διαπραγματευόμαστε χωριστά με αυτές τις χώρες. Και αυτό μπορεί ε, τοποθετεί μάλλον ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μειονεκτική θέση. Υπάρχουν ε, δυσανάλογες συμφωνίες και από αυτές οι χώρες πολλές φορές κατηγορούν την Ευρώπη πως υποφελείται από διμερείς συμφωνίες. Και αυτό μπορεί να επιβαρύνει τις οικονομικές σχέσεις με αυτέ τι χώρε. Και έπειτα υπάρχουν ακόμα δύο αίτια που τα οποία πρέπει να αξιολογήσουμε. Είπατε κύριε Βέμπερ ότι τα προβλήματα της Ανατολικής Ευρώπης είναι σημαντικά επίσης, χωρίς αμφιβολία. Αλλά η εντύπωση που έχω τα τελευταία χρόνια είναι πως η Ευρώπη συνολικά έχει μετακινήσει τα ενδιαφέροντά της προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη και όχι προς την Μεσόγειο. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο των οικονομικών πόρων, αλλά και της δυνατότητας να παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν. Και καταλήγω με την τελευταία μου παρατήρηση. Η Ευρώπη βασικά έχει στραφεί προς αυτές τις δύο χώρες και έχει βασιστεί σε δύο θέματα. Τρομο, Ισλαμική τρομοκρατία και το θέμα της μετανάστευσης. Και από αυτού βασίσαμε τις υποθέσεις χρηματοδότησης, την τεχνική βοήθεια, κάποιες μετριοπαθείς πολιτικές πιέσεις προς αυτές τις χώρες και όλα όσα κάναμε μας έδειξαν και αποδείχτηκαν μάλλον ωφέλιμα στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Αλλά εδώ δεν λειτουργούν και δεν λειτουργούν γιατί υπάρχει έλλειψη οράματος, μακρόπνοου οράματος. Υπάρχουν ε, Υπάρχει δυσπιστία και υπάρχει και ανεπάρκεια των πόρων. Και αυτό υπόθηκε όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία. Και όλα αυτά επιδρούν αρνητικά. Και εγώ θέλω να τονίσω γιατί πρέπει να προσέξουμε γιατί όλα αυτά τα προβλήματα μπορεί αρνητικά να επηρεάσουν και πολύ έντονα. Σε πρόσφατη μου επίσκεψη που έκανα στη Μαυριτανία το είδα να αποδεικνύεται στην πράξη και έχω μια ερώτηση κλασική. Ίσως θα ήταν καλύτερο η, το πιο τομεακές παρεμβάσεις να έχουν ένα όραμα πιο μακρόπνο. Εσείς ε, παρενέβετε σε θέματα οικονομικά, αλλά κυρίως θα πρέπει να μας ασχολήσει η πολιτική στάση και η θεσμική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μιλανμόν. Ευχαριστώ πάρα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σας ενώπιόν μας σήμερα που μας μιλάτε για μια τόσο σημαντική περιοχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι και για τις ε, χώρες της Βόρειας Όχθης της Μεσογείου και είναι και η περίπτωσή μου. Ισπανός είμαι, δεν χρειάζεται να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η περιοχή για όλους εμάς. Ο κύριο Παντζέρη είπε πολλά πράγματα και ε, μα κάλυψε όλου, δεν θα μακρηγορήσω. Βασικά δύο ερωτήσει έχω να σα κάνω. Το θέμα τη γραμματεία, στο οποίο αναφερθήκατε και οι δυο σα. Τι προβλήματα ελπίζετε ή περιμένετε να λύσει η γραμματεία αυτή. Δηλαδή, Ποια θα είναι τα ευεργετήματα της γραμματής αυτή που δυστυχώς ακόμα δεν λέω ότι είναι σε εμπλοκή αλλά κάπως σε κάποια δυστοκία. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία που περιμένετε και ελπίζετε. Ο κύριος Βέμπερ κάποια στιγμή είπε ότι είναι απολύτως απαραίτητη. Αλλά διείδα και κάποια επιφύλαξη για το πώς θα λειτουργήσει αποτελεσματικά. Παραμένω, κρατώ αυτό που είπατε, ότι είναι απολύτω απαραίτητη, αλλά μπορείτε λίγο να επεκταθείτε στην αναγκαιότητα αυτή. Και ε, ένα δεύτερο, είπατε και εσείς και ο κύριος Φοντέν την ανάγκη να προωθηθεί η περιφερειακή συνεργασία, δηλαδή η συνεργασία νότου-νότου, για να ε, τραβήξουν περισσότερες επενδύσεις, να προσελκύσουν. Βεβαίως είναι αυτό οπωσδήποτε ε, απαραίτητο. Έχουμε όμως μια μεγάλη επιφύλαξη. Ε, πού είναι ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος νότου-νότου. Βλέπουμε πόσο κλειστά είναι αδιαπέραστα τα σύνορα σχεδόν Αλγερίας-Μαρόκου. Εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε από το βορρά για να γίνει πραγματικότητα και να μην είναι χήμερα η συνεργασία αυτή νότου-νότου. Κυρία Μπέναραμπ. Ε, euh, Σας ευχαριστώ ζούμε μια ενεργειακή και άλλη κρίση και επομένως η ευρωμεσογειακή ζώνη είναι απαραίτητο να βγει από την εξάρτηση στα ορυκτά καύσιμα και να χρησιμοποιήσει τις ανανεώσιμες πηγές. Το δράμα του Τσερνομπίλ και οι επιπτώσεις του στην υγεία των πληθυσμών γύρω από εκεί δείχνει ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι καθαρή ενέργεια ούτε ανανεώσιμη. Επειδή εξάλλου η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας μπορεί εύκολα να τύχει κατάχρησης προς τη στρατιωτική χρήση και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα από τη στάση του Ισραήλ που διαθέτει το πυρηνικό όπλο και δεν έχει συνυπογράψει τη συνθήκη μη διάδοσης. Για όλους αυτούς τους λόγους σήμερα δηλώνουμε ότι η μόνη λύση για να υπάρξει αποκλιμάκωση στην ανάπτυξη των πυρηνικών είναι ότι επειδή οι χώρες λοιπόν που δεν έχουν τον, πυρηνικό, τον πυρηνικό όπλο θα θελήσουν σύντομα το Πουτίν, η μόνη λύση επαναλαμβάνω είναι στην ευρωμεσογειακή ζώνη να υπάρξει πλήρης αποπυρηνικοποίηση. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Γαλλία συνεχίσει να πωλεί αυτή την τεχνολογία τότε οδηγούμαστε προς την καταστροφή και θα καταλήξουμε στη δημιουργία τεραστίων αποθεμάτων καρκινογόνων πυρηνικών αποθεμάτων. Τα παιδιά μας θα μας κατηγορήσουν και θα έχουν δίκιο, αλλά θα είναι πολύ αργά. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να βγούμε από την πυρηνική ενέργεια. Ποια χρηματοδότηση υπάρχει για τη χρήση ανανεωσίμων πηγών ενεργείας στα πλαίσια της Ένωσης για τη Μεσόγειο και τι σχέδια έχουν ήδη προβλεφθεί. Σας κατευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μαριέλ Ντεσαρνέζ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να επανέλθω σε αυτό το θέμα της ενέργειας, ίσως από κάποια διαφορετική έποψη. Η κοινή διαχείριση των υδάτων για τις χώρες αυτές του Νότου είναι κάτι το πρωτεύον διότι μπορεί έτσι σε πολιτικό επίπεδο να δημιουργηθούν συμμαχίες που δεν θα δημιουργούνταν αλλιώ στο καθαρά πολιτικό επίπεδο το ενεργειακό θέμα είναι ουσιώδες και επομένως θα ήθελα να μου πείτε και οι δύο τι φρονείτε για την επιχείρηση Desertec. Πρόκειται για εκατοντάδες εκατομμυρίων νερό για τη δημιουργία τεραστίων εκτάσεων ηλιακών συσσωρευτών στην έρημο. Το θέμα αυτό είναι καθα... μεγάλης πολιτικής σημασίας, θέτει το πρόβλημα της χρηματοδότησής του αλλά και της φιλοσοφίας του. Υπάρχουν επενδυτές, για να το πω έτσι γενικά, Ευρωπαίοι ώστε να δημιουργηθεί η ηλιακή αυτή ενέργεια ενέργεια και να μεταφερθεί μετά στην Ευρώπη ή μήπως υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί χρηματοδότηση νότου-νότου ή λιγότερο κερδοφόρα για να το πω έτσι επίσης επένδυση ώστε αυτή η τεράστια επιχείρηση Tech να ωφελήσει όντως τους κατοίκους του νοτιού τμήματος της Μεσογείου κυρίως και όχι κυρίως στην τροφοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση, συνάδελφος Γιαννάκου και μετά και πάλι ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας ακρόασης καθώς και τα, σχόλια για τις επιτυχίες, πιθανές επιτυχίες ή αποτυχίες. Ε, έχω την εντύπωση ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι αν πραγματικά έχει γίνει αξιολόγηση των μέχρι σήμερα υπαρχόντων προγραμμάτων. Ουσιαστική αξιολόγηση για την πραγματική τους επιτυχία ή αποτυχία. Και η επιτυχία ή η αποτυχία τους πρέπει να δούμε πού απευθύνεται. Δηλαδή τα προγράμματα αυτά γίνονται με στόχο ε, για να, επιστραφούν όλα τα χρήματα στις μεγάλες τεχνικές εταιρείες που κάνουν τα διάφορα έργα. Οπότε επιστρέφονται σε εταιρείε συγκεκριμένων χωρών, μεγάλων χωρών της Ένωσης ή ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε πραγματικά τις χώρες αυτές. Και το ερώτημα είναι, τις βοηθάμε όταν τα ζητήματα της δημοκρατικής διακυβέρνησης, της ε, συμμετοχής όλων των πολιτών και της συμμετοχής των γυναικών παραμένουν στο περιθώριο της ευρωμεσογειακής αντίληψης. Ε, εγώ έχω την εντύπωση κύριε Πρόεδρε και θέλω να ρωτήσω τους ε, συμβάλλοντες σήμερα σε αυτή τη συζήτηση Έχω την εντύπωση ότι η βοήθεια προς τις οποιασδήποτε χώρες του κόσμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνονται με βάση ρήτρε και προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις είναι να μην συμμετέχουν οι κυβερνήσεις που στην ουσία χρηματοδοτούνται στο οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο ναρκωτικών και να συμβάλλουν στην εξέλιξη της δημοκρατίας η οποία εξέλιξη της δημοκρατίας και στη Μεσόγειο και στον Ισλαμικό κόσμο δεν είναι αυτή που νομίζουμε που πρέπει να είναι στην εποχή μας. Η δε κατάσταση επί της ουσίας στις χώρες αυτές, παραδείγματο χάρη στην Αίγυπτο, όταν επί 1436 ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κολεγίων και πανεπιστημίων, μόνο τα 30 χρηματοδοτούνται από το κράτος και τα υπόλοιπα από Ισλαμικές οργανώσεις, υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Τι θέλουμε πραγματικά να κάνουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε ή και αν μου επιτραπεί να πιέσουμε τις χώρες αυτές προς τον εκδημοκρατισμό. Ή αυτό δεν μας ενδιαφέρει τελικά και αυτό που είναι ουσιαστικό είναι μόνο business και οικονομικές παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Eh, να ρωτήσω τον εισηγητή αν θέλει να παρεμβεί τώρα ή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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την τελευταία παρατηρήση. Μόλις τελειώνουν 18 μήνες αξιολόγησης. Με την έκθεση των συμβούλων που μας αξιολόγησαν υπό το καλοσυνάτο βλέμμα <laughs> της Επιτροπής, που όμως ε, κάποιε φορές είναι και επικριτικό, μαζί με την Επιτροπή των Σοφών έχετε όλα τα στοιχεία για να λάβετε τι πολιτικέ αποφάσει που πρέπει να λάβετε και του προσανατολισμού που θέλετε να μα ε, δώσετε. Έχετε δηλαδή αυτό το σημαντικό σημαντικό, τη σημαντική τεκμηρίωση που είναι στη διάθεσή σα. Δεύτερη παρατήρηση για την απαραίτητη περιφερειοποίηση που σας είπα πριν από λίγο για την συνεργασία νότου-νότου. Πιστεύω πως αυτό είναι απαραίτητο στο πρόγραμμά μας και σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ότι δηλαδή ένας ε, ε, Αιγυπτίος φορέας έφτιαξε την πρώτη τσιμετοβιομηχανία στην Αλγερία είναι την ίση, οι οποίοι εξάγουν, επίσης υπάρχουν την και εταιρείε που προσπαθούν να βγάλουν προς το Μαρόκο και την Αλγερία την ε, δική τους ε, χρημα, ε, χρηματοπιστωτική τεχνογνωσία. Άρα λοιπόν εκεί γίνεται η συνεργασία στο τομέα του ηλεκτρισμού και είμαι στην φάση υπογραφής με την Παλαιστινική Αρχή από τη μια πλευρά και λίγους μήνες αργότερα με την αντίστοιχη αρχή από την ε, Ισραηλινή πλευρά ε, και όταν μιλώ για συνεργασία, για περιφερειοποίηση είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία κάποια στιγμή μπορεί βέβαια να ε, συμβολιστούν με μεγάλα έργα υποδομής αλλά που καθημερινή, στην καθημερινή λειτουργία τους ε, αφορούν την ε, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Τώρα για την ενέργεια και το κλιματικέ τις κλιματικές αλλαγές. Πιστεύω ότι για να δώσουμε νόημα στην παρέμβασή μας στα νότια παράλια της Μεσογείου είναι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα δείτε ότι η έκθεση Κονσουή προτείνει τα 2 δις ευρώ που είχαν μπει στο αποθηματικό στην διάμεση αναθεώρηση των εντολών που είχε λάβει η ΕΤΕ προτείνουν να αφιερωθεί το σύνολο αυτών των 2 σε αυτόν το τομέα, την καταπολέμηση δηλαδή των κλιματικών αλλαγών και τις απαραίτητες προσαρμογές στον ενεργειακό τομέα και αυτό συγκεντρώνει τη δική μας ε, σύμφωνη γνώμη, αλλά εσείς θα το αποφασίσετε. Αυτό τι σημαίνει δεν σημαίνει μία τεχνολογική πρόκληση. Εγώ δεν θα εκφραστώ όσον αφορά το θέματα ασφάλειας ε, της ε, πυρηνικής ενέργειας, γιατί αυτά ξεπερνούν τις αρμοδιότητες της ΕΤΕ, αλλά αυτό σημαίνει πως ίσως αύριο μεθαύριο χρειαστεί να χρηματοδοτήσουμε ένα πυρηνικό σταθμό στην... Ε, στην υπεριορδανία. Άρα λοιπόν, κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη της δικής, της του ενεργειακού μείγματος, γιατί να το απαγορέψουμε αυτό στις χώρες του Νότου, ενώ αυτό γίνεται στην, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ΕΤΕ υιοθετήσαμε την ίδια πολιτική για τον Νότο, όπως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, κάθε κυρίαρχο κράτος θα αποφασίσει τη δική του ενεργειακή προμήθεια, ανεφοδιασμό. Και αυτό και ενθαρρύνουμε τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θέτουμε πολύ φιλόδοξο στόχο στόχους. Τώρα το πρόγραμμα Desertec, Desertec που το αναφέρατε πριν από λίγο κυρία Ντεσαρνές είναι κάτι πολύ μακροπρόθεσμο όπως στην πράξη είναι ένα ηλιακό μεσογειακό πρόγραμμα στο τετράγωνο. Εγώ κάλεσα στο Λουξεμβούργο το σύνολο των συμβαλωμένων μερών στο Desert ώστε να μην προσπαθήσουμε να φέρουμε σε αντίθεση τις διάφορες τεχνολογίες. Αυτό θέτει πολύ σημαντικά προβλήματα. Έχουμε αναφερθεί κατά στο θέμα του νερού. Αν έχουμε χιλιόμετρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα φωτοβολταϊκών επιφανειών θα πρέπει να μπορούμε και να τις καθαρίσουμε για να είναι αποτελεσματικές. Επίση, θα πρέπει να αυξηθεί η δυνατότητα εξαγωγή ενέργεια από την νότια όχθη της Μεσογείου προς την Ευρώπη. Δηλαδή θα πρέπει να καταστεί οικονομικά βιώσιμο ένα πρόγραμμα παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια με βάση την ε, ηλιακή ενέργεια, που δεν θα ήταν βιώσιμο στην Νότια Μεσόγειο, γιατί τιμέ ηλεκτρισμού που οι καταναλωτέ είναι έτοιμοι να πληρώσουν στο σύνολο των χωρών τη Νότια Μεσογείου πέρα από το Ισραήλ είναι πολύ χαμηλότερε από, ε, από το επίπεδο σκοπιμότητας ε, που αφορά αυτό το πρόγραμμα ηλιακής ενέργειας. Και έτσι ολοκληρώνω. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών. Συνάδελφοι, συγγνώμη, διακόπτει ο Πρόεδρος ησυχία ε, από σεβασμό προς τον ε, ομιλητή και τον εισηγητή η χώρα η οποία ηγείται του προγράμματος είναι το Μαρόκο που μόλις δημιούργησε ένα νέο οργανισμό που είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στην ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας και εδώ έχουμε ολοκληρώσει τη σύναψη μιας εταιρικής σχέσης με τον οργανισμό αυτό ώστε να μεταφέρουμε αυτές τις τεχνολογίες και να καταστούν βιώσιμες οι επενδύσεις αυτές. Πρόεδρε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός. Λοιπόν, για τις κλιματολογικές αλλαγές αλλά και για τα ερώτημα της κυρίας Ντεσαρνές, της κυρίας Μπεναράμπ και των υπολείπων για τις ανανεώσιμες ενέργειες, το περιβάλλον και το ξαναλέω τις κλιματολογικές αλλαγές. Ένας από τους κύριους άξονες ανάπτυξης των προγραμμάτων της Ένωσης για τη Μεσόγειο είναι ακριβώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο περιβάλλον. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες αλλά και δυνατότητες επίσης τεράστιες. Καλό είναι να γίνεται κανείς ε, ευεργέτης και δωρητής, αλλά επίσης καλό είναι να γνωρίζουμε ότι πρόκειται και για μια τεράστια αγορά όπου μπορούν να αναπτυχθούν οι δραστηριότητε και των ευρωπαϊκών εταιριών και των ε, μεσογειακών εταιριών σε εταιρικό σχέση. Μπορούν λοιπόν να υποφεληθούν οι επιχειρήσεις και να γίνουν τεχνολογικές προοδοί με όλα αυτά τα προγράμματα. Γι' αυτόν τον λόγο το συνδέω αυτό που είπαμε, με αυτά που είπε και ο κύριος Παντζέρη. Δεν πρέπει να φοβηθούμε μήπως ορισμένες χώρες μέλη παραγνωρίσουν τις χώρες του Νότου της Μεσογείου και ενδιαφερθούν μόνο για τις Ανατολικές. Διότι ακριβώς στην Ένωση οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε βρίσκονται και στο Νότο και στην Ανατολή και όλα συνδέονται οι μεταναστευτικές ροές, η ενέργεια, το κλίμα, όλα αυτά δεν έχουν σύνορα. Και όταν, αφού οι οικονομίες μας συνδέονται όλες, ας μην τις αναφέρω μία-μία, αφού λοιπόν υπάρχει μια τέτοια αλληλεξάρτηση ενεργειακή, βιομηχανική, στις υπηρεσίες οικονομική, στρατηγική και περιβαλλοντολογική γι' αυτόν τον λόγο θα ήταν αφελής και όποιος θα νόμιζε ότι επειδή βρίσκεται στο βορρά μπορεί να πάψει να ενδιαφέρεται για το νότο ή το αντίθετο. Όλα συνδέονται, το μέλλον μας εξαρτάται τον μεν από τους δε. Και το θέμα της Μεσογείου επομένω ενδιαφέρει και τις νότιες χώρες και τη Γερμανία και τις άλλες βόρειες χώρες. Και το ίδιο ισχύει και για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτή είναι ακριβώς η φιλοσοφία της πολιτικής της καλής γειτονίας. Η οικονομική σταθερότητα πρέπει να υπάρξει και στον Νότο και στην Ανατολή. Η κυρία Γιαννάκου είχε πει ότι η αποτίμηση των υπαρχών, για την αποτίμηση των υπαρχών προγραμμάτων σας διαβεβαιώνω ότι όλα αυτά τα προγράμματα και τις ΕΤΕ και τα υπόλοιπα την χάνουν μιας περιοδικής και κατά τακτά χρονικά διαστήματα αξιολόγησης που γίνεται γνωστή και από το Κοινοβούλιο και δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα, στη σχετική ιστοσελίδα. Δεν επηρεάζονται οι μελέτες, οι αξιολογήσεις αυτές από τίποτα. Τώρα, στις μεσογειακές χώρες ίσως δεν είναι ότι έχει γίνει τέλειο, αλλά τα αποτελέσματα της ευρωμεσογειακής πολιτικής και της διαδικασίας της Βαρκελόνης διότι δεν είναι αρνητικά διότι μπορώ να σας πω ως άνθρωπος που συνεργάζεται από το 90 και μετά με, στην επεξεργασία των μεσογειακών θεμάτων μπορώ να σας πω ότι είναι πολύ εύκολες οι επικρίσεις αλλά κατ' εμέ η διαδικασία της Βαρκελόνης είναι επιτυχία Βέβαια όλα εξαρτώνται από τους στόχους που έχουμε καθορίσει. Αν κάποιος φανταζόταν ότι η διαδικασία της Βαρκελόνης θα επέτρεπε την ειρήνευση της Μέσης Ανατολής, τότε είναι αποτυχία. Αλλά θα έπρεπε κανείς να είναι αφελής για να πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνευση από μια οικονομική απλή απλώς διαδικασία όπως της Βαρκελόνης. Μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση κάποιου διαλόγου, αλλά γενικά και για τα, τις τρεις πτυχές που αναφέραμε είναι αυτά τα αποτελέσματα της διαδικασίας της Βαρκελόνης. Και στο βορρά και στο νότο και στην Ανατολή ισχύουν ανάλογα κριτήρια. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και με αυτά τα ρεαλιστικά κριτήρια η Βαρκελόνη είναι επιτυχία. Ίσως να έπρεπε να προχωρήσει περαιτέρω, δεν λέω. Τώρα για τη γραμματεία, γιατί είναι απαραίτητη, μα αυτό προκύπτει από όλα όσα είπα η γραμματεία είναι απαραίτητη διό, για να υπάρχει ως ένας χώρος όπου συγκεντρώνονται, συνεννοούνται όλοι. Όλοι οι εταίροι της Ένωσης για τη Μεσόγειο συνεννοούνται σε επίπεδο βέβαια υπουργικό, αλλά εκεί δεν υπάρχει καμία συνέχεια για την Ένωση για τη Μεσόγειο. Η γραμματεία της θα αποτελούσε ακριβώς αυτόν τον κοινό για όλους τόπο όπου θα γίνεται ο συντονισμός και ο συνδυασμός και η συνεννόηση και η διαχείριση βέβαια, η δημοσιονομική η χρηματική διαχείριση όλων των προγραμμάτων. Τελεία. Ωραία, σας ευχαριστώ. Μια τελευταία ώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Πεγιόν για να ε, συνοψίσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρο, ευχαριστώ συνάδελφοι για τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις και τα ε, σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ και τους δύο μιλητές για τις αναλύσεις σας. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με τρεις παρατηρήσεις για τα όσα με βάση τα όσα είπε ο φίλος και συνάδελφος Πανζέρη. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να ρισκάρουμε την αποτυχία και γι' αυτό και θα πρέπει έντονα να εκδηλώσουμε τη βούληση του Ευρωκοινοβουλίου να συνοδεύσει και να εμπλακεί στη διαδικασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Είναι μια οικονομική πρόκληση, γεωστρατηγική πρόκληση, αλλά και πολιτιστική. Και μια Ευρώπη η οποία είναι κλεισμένη στον εαυτό της και που ασχολείται με τον Νότο μόνο μέσω της μετανάστευσης και του φόβου είναι μια Ευρώπη που δεν είναι σε θέση να παίξει ρόλο της στην παγκοσμιοποίηση. Και δεν θα ήθελα η κατάσταση και η οχλαγωγία που επικρατεί εδώ μέσα κατά τη διάρκεια αυτής της ακρόασης ε, και οι διαφωνίες που ακούγονται από δεξιά και αριστερά θα πρέπει να σας κάνουν να αμφισβητήσετε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου ως προς το θέμα. Και έπειτα μιλήσατε για τη Γενική Γραμματεία. Όσοι ε, νοιάζονται για την διαδικασία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να διαπιστώσουν πως μόνο μέσα σε αυτή τη Γενική Γραμματεία βλέπουμε να κάθονται στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων Ισραηλινοί με Παλαιστίνιους. Και ε, εντάξει, μπορεί κανείς να στραβομοτσουνιάζει, αλλά μπορεί και να χαιρετίζει τις σημαντικές πρόοδους. Και από εκεί και πέρα πιστεύω πως η φιλοσοφία μας, αυτή που θέλουμε να υιοθετήσουμε και έχω μάλιστα σημειώσει ότι ο Παλαιστίνιος Πρωθυπουργό και βασίζομαι στα στοιχεία τα οποία μα δώσατε, χαιρετίζει την πολιτική συγκεκριμένων προγραμμάτων ω προετοιμασία για την ειρήνη και στα κατεχόμενα. Πιστεύω λοιπόν ότι το να προχωρήσει το πρόγραμμα τη Ένωση για την Μεσόγειο μέσα στο θεσμικό πλαίσιο το σημερινό είναι ένα από τα στοιχεία που θα μας επιτρέψει και τόσο το καλύτερο αν η Ευρώπη πάρει την πρωτοβουλία γι' αυτό θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε προς μια λύση. Τρίτη παρατήρηση αγαπητοί συνάδελφοι είναι πως θα υπάρξει μια, ένα θέμα που δεν μπορούμε να το λύσουμε σήμερα αλλά που θα το έχουμε να το αντιμετωπίσουμε στη συζήτησή μας που θα αφορά την θεσμική και δημοκρατική διοργάνωση για τους βουλευτές της Ένωσης δηλαδή μια γενική γραμματεία πολύ ωραία και καλά ε, Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξης υπέροχα, η Κομισιόν, τα κράτη και ναι, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σήμερα το θέμα αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί πώς εμείς θα μπορέσουμε όχι μόνο, μόνο το ότι είμαστε, λόγω του ότι είμαστε δημοσιονομική αρχή, αλλά και με την παρουσία μας πώς θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τα προγράμματα, να, κάνουμε την αξιολόγησή μας και να συμμετέχουμε στις συζητήσεις όπου το επιθυμούμε. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε με την κινητοποίηση της ε, κοινωνίας των πολιτών, με τις ε, περιφέρειες. Ε, θα πρέπει και το Ευρωκοινοβούλιο, όχι από καιρού καιρών και όχι μόνο σε σχέση με την την δημοσιονομική πολιτική, αλλά για το σύνολο τη παρακολούθηση των προγραμμάτων και τη συνεργασία να συνεργάζεται, γιατί αυτό είναι και το πνεύμα τη Ένωση για τη Μεσόγειο, σε συνεργασία με του συναδέλφου βουλευτές του Νότου, τη άλλη όχθη. Και εδώ αυτό θα πρέπει να μα απασχολήσει. Σα ευχαριστώ και του δύο για τις, ε, τα στοιχεία που μα δώσατε σήμερα. Σα ευχαριστώ και εγώ για την εξαιρετική σας ε, παρουσία και κλείνουν οι εργασίες εδώ. Bene Ωραία, συνάδελφοι παρακαλώ, όσοι θέλουν να μπουν ή να βγουν από την αίθουσα να το πράξουν σύντομα παρακαλώ, γιατί έχουμε διάφορες εκθέσεις, θα ψηφίσουμε πολλές τροπολογίες και έπειτα ακολουθεί το διευρυμένο προεδρείο, όπως πάντα δηλαδή, είμαστε με το χρόνο μετρημένο. Θα ήθελα να τοποθετήσετε την ηλεκτρονική σας κάρτα στην κατάλληλη σχίσμη, ώστε να κάνουμε μία δοκιμή. Να κάνουμε δοκιμή ή να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε και το βλέπουμε στην πορεία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το σχέδιο γνωμοδότησης που φέρει την υπογραφή της κυρίας Λοκ Μπίλερ. Είμαστε στην τροπολογία άρθρο 1.1. Τροπολογία 4. Και 22 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 23. Τη εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται προφορική τροπολογία τη συντάκτρια. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υποσύρεται 7 και πάμε στην 24 τη ηγητρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Όπω πάντα δεν ρωτώ τι εποχέ. Αν θέλει κάποιο να απέχει να μου το πει. 8 τη εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 25. Της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχέ... Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Μήπως να κάνουμε μπλοκ. 16, 17 και 18 συμφωνείτε. Υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 19 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 28 υπέρ κατά απορρίπτεται στο πάμε στην 21 υπέρ κατά εγκρίνεται 2 είναι το εκτιμώντας 5 υπέρ κατά εγκρίνεται η 3 τώρα στο εκτιμώντας 6 της εισηγητρίας υπέρ κατά εγκρίνεται Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης, όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Περιμένω να ψηφίσετε όλοι. Άντε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Νομίζω πως ψήφισαν όλοι. Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 57 υπέρ, 1 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται συγχαρτήρια στην εισηγήτρια. Τώρα, περνάμε στο σχέδιο έκθεσης όπου η συγκητής είναι ο συνάδελφος Ντανζόν. Παράγραφος 1, τροπολογία 5. Λέζινγκ, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 6, κόπα Πάσκου, γκουαλτιέρι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 7. Μπουτικόφερ Μπράτνερ υπέρ κατά εγκρίνεται. 8. Γιάννε Μπαρνουέβο Γκαρσία υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά απο, εγκρίνεται. 9. Λέζινγκ υπέρ κατά απορρίπτεται. Ναι. Συμβιβαστική 1 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 12 γιατί οι υπόλοιπε καταπέπτουν. Γκόμε υπέρ κατά απορρίπτεται. 13. Κοπά Πασκού Γκολτιέρη υπέρ κατά εγκρίνεται. 14. Κοπά Πασκού Γκολτιέρη υπέρ κατά εγκρίνεται. 15. Οι ίδιοι συγητές υπέρ κατά εγκρίνεται 16 υπέρ κατά εγκρίνεται προφορική τροπολογία Κόβαλ Βανόρδεν υπέρ κατά απορρίπτεται <clears throat> περνάμε στη συμβιβαστική 2 του εισηγητή υπέρ κατά αποχε, ε, συγγνώμη, εγκρίνεται Πάμε στην 24 παράγραφος 5α. Είναι τρία διαφορετικά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Δεύτερο, ε, τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 25. Μπουτικόφερ Μπράτνερ υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 26 Van Orden υπέρ κατά απορρίπτεται 27 Μποτικόφερ Μπράτνερ ε, υπέρ κατά εγκρίνεται προφορική τροπολογία 3 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται πάμε στην 29 Κέλαμ υπέρ κατά εγκρίνεται 30 Γιάννα Μπαρνόεβο Καρσία υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. 31. Νταφ. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το πρώτο τμήμα της 31. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Chiudiamo la votazione. Τέλος της ψηφοφορίας. 29 κατά 33 υπέρ εγκρίνεται με μία αποχή. Τρίτο τμήμα του, της τοπολογίας 31, λέει ο, ο πρόεδρος. Ζητά συγγνώμη και διορθώνει δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 32 πανόρντεν υπέρ κατά απορρίπτεται 33 νταφ υπέρ κατά απορρίπτεται 34 υπέρ κατά α, εκρίνεται. 35 υπέρ κατά Εκρίνεται. 36 υπέρ κατά Εκρίνεται. 37 υπέρ Α, δεν την ψηφίζουμε γιατί είναι ταυτόσιμη με 36 όπως είναι και γραμμένο και στις σημειώσεις. Λοιπόν, 38 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 του εισηγητή υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 46 γκάλερ υπέρ. Κατά. Άμα δεν σηκώνετε τα χέρια σας, δύσκολο να δούμε τι... Ας τα ξανακάνουμε. Λοιπόν, 46 υπέρ... Α, εντάξει, τώρα κατάλαβα. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Πολύ ωραία τα πάτε, μπράβο. Κατά, εγκρίνεται. 48 υπέρ. Α, υπέροχα. Έβγε σε όλους απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 31, δύο τμήματα. Α, όχι. Έκανα λάθος σελίδα. 52. Ναι, είχα διπλώσει λάθος σελίδα μου. Λοιπόν, 52 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά εγκρίνεται. 54 άντε για την 53 ωραία. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 53 γκάλερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Chiudiamo? No, ancora qualcuno. 33 contrari, 31. Απορρίπτεται. 31-33. 54. Ή 54 ψήφι Κατά. Απορρίπτεται. Ή 55 είπε. Κατά. Απορρίπτεται. 56 είπε. Κατά. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 58 υπέρ. Ε, Κατά. Απορρίπτεται. 59 Επέ. Κατά. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η προφορική υπαριθμών 4 του εισηγητού ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 62. Ψήφι Κατά. Απορρίπτεται. 63 Επέ κατά απορρίπτεται 64 υπέρ κατά απορρίπτεται 65 υπέρ κατά απορρίπτεται 66 υπέρ ο κύριος Νταφ παρακαλώ να γίνει έλεγχος για την 65 γιατί εγώ νομίζω ότι εγκρίθηκε. Απροβάτο, όχι ρεσπίντο. Όχι, ρε Σπίντο. Αφού είπαμε ότι έχει απορριφθεί. Νομίζω ότι ήταν σαφές άλλωστε. Μα την έχουμε ήδη ψηφίσει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να επανέλθουμε. Εγώ νόμιζα ότι ήταν σαφής η απόρριψη. Ρωτάω τη γραμματεία. Τι γίνεται τώρα. Έχουμε αποφανθεί. Μπορούμε να την ξαναψηφίσουμε. Τι διαδικαστικό υπάρχει. Εγκρίνεται ο έλεγχος. Εντάξει. Ωραία. Ας ψηφίσουμε τότε ηλεκτρονικά την 65 παρακαλώ. Ονομαστικά, ηλεκτρονικά, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 65. Chiudiamo la votazione. Πέρασε. 52 κατά, ε, μάλλον απερίφθη, ξέρω εγώ. In pace, onorevole Duff. 66. Eh. Εντάξει, κύριε Ντάφ, εισχάσατε. 66 είπε κατά απορρίπτεται. 67 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτον ψήφι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Το 68 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η 69 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. Η 71 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 72 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 73 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 74 υπέρ κατά απορρίπτεται 75 δεν ψηφίζεται 76 υπέρ κατά απορρίπτεται 77 υπέρ κατά απορρίπτεται 78 υπέρ κατά απορρίπτεται 79 υπέρ κατά απορρίπτεται 80 υπέρ κατά απορρίπτεται 81 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η προφορική υπαριθμών 5 του εισηγητή ψήφι υπέρ κατά εγκρίνεται. Η συμβιβαστική τώρα υπαριθμών 4 ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά εγκρίνεται. Άρα θα πρέπει να πάμε τώρα στην 94 ψήφι υπέρ. Κατά απορρίπτεται 95. Α, καταπίπτει sì, sì, sì, certo, certo. Α, τσεκ θέλετε. Καλά. Τι favorevoli. 96 υπέρ κατά. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ε, έχετε χαλαρώσει, δεν θέλετε να σηκώνετε χέρια. 99 υπέρ. Ε, ευχαριστώ. Κατά, εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Απορρίφτεται. Η προφορική υπαριθμό είναι 9 του εισηγητή ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 103 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προφορική του συγητή 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα τώρα θα πρέπει να πάμε στην 105 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ακολουθεί τώρα block. 106, 110, 113, 115. Ψήφι υπέρ παρακαλώ κατά απορρίπτεται 107 υπέρ κατά απορρίπτεται 108 υπέρ κατά απορρίπτεται 109 υπέρ κατά εγκρίνεται 111 υπέρ Α, όχι, πρέπει να πάμε σε 114, τι λέτε. Όχι, για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα. 111. Ο κύριος Νταφ. Η γκόμε, η 109 εγκρίθηκε, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, για να το διευκρινίσω, δεν έχω καμία αμφιβολία. Απρομπάτο είπα, εγκρίνεται. Ορίστε. Για το 111 δεν κατάλαβα ποια ήταν η αντίδρασή σας. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 111, ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 11 προφορική του εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η προφορική 12 του εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η προφορική πάντα 13 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ορίστε. Ο κύριος Λάμστορφ, παρακαλώ. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε. Κατά κανόνα, όταν ψηφίζουν μαζί οι πράσινοι, ε, σοσιαλιστές και φιλελεύθεροι, εσείς ε, αποκεκτημένοι ταχύτητα λέτε ρησπίν, το απορρίπτετε. Δύο φορές σας έχει συμβεί, δεν θέλουμε να ζητάμε παλήθευση κάθε φορά. Αλλά τι θα γίνει τώρα. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την, την προφορική 13. Τώρα δεν ξέρω ποια τροπολογία ήταν καν, αλλά ήταν πάλι μια ψηφοφορία όπου όλη αυτή η πτέρυγα ψήφισε υπέρ και ακούτε μετά ρεσπίν το να λέτε. Όταν ψηφίζουν πράσινοι σοσιαλιστές και φιλελεύθεροι εγκρίνεται η τροπολογία. Non ε, Ούτε εγώ δεν θυμάμαι τώρα τι θα γίνει. Θέλετε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την προφορική 13. Καλώ. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την προφορική 13. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρα. 31 κατά, 33 υπέρ, 0 αποχές, μάλιστα Ε, όταν υπάρχουν αυτές οι μικρές διαφορές στην ψηφοφορία, αν δεν σηκώνετε χέρια, εγώ πώς να σας μετρήσω. Τι να κάνω. Α, υπήρχε ένας Ιταλό ηθοποιό, Πέτρο Λίβι το λέγανε, που συχνά όταν εκείνος μιλούσε, ε, άκουγε τους ακροατές, τους θεατές μάλλον και του φωνάζανε αυτοί, αυτοί ότι δεν ακούγανε και εκείνος τότε τους φώναζε βότσε, φωνή. Ε, και, πήγαινε, και πήγαινε λέγοντας η ιστορία. Λοιπόν, την 115 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 117 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ωραία. 118 ε, υπέρ, κατά. Ωραία, τώρα σας βλέπω καλά. Απορρίπτεται. 119 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 120. Όπως και η ίδια με την προηγούμενη. 121. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 122 και 125 μπλοκ υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 123 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα του 123. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 34 κατά, 30 υπέρ, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της 123 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 124 υπέρ, κατά εγκρίνεται 126 υπέρ κατά απορρίπτεται 127 υπέρ κατά απορρίπτεται 128 υπέρ κατά απορρίπτεται 129 υπέρ κατά, απορρίπτεται 130 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Όχι, πρόεδρε, συγγνώμη. Κάποιο διακόπτη. Δεν βλέπουμε ποιο είναι. Μου επιτρέπετε. Εγώ θέλω να αποσύρω την 132 και τη 232 και τη 233. Γιατί καλύπτονται από άλλες τροπολογίες. Bene, allora 132 lo saltiamo e poi Ωραία λοιπόν, την 132 την αφήνουμε, 133 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται, 134 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 135 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Ε, εντάξει, εντάξει. Ε, να ψηφίσουμε για το δεύτερο τμήμα του 135. Τέλος ψηφοφορίας. 36 υπέρ, 24 κατά. Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Απο... Εγκρίνεται. 139 καταπίπτει. Πάμε στην 140 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 14. Του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 15 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στο 150 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. <clears throat> Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά εκρινέται 156 υπέρ κατά, κατά. απορρίπτεται 157 υπέρ, Κατά. Απορρίπτεται 158 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 159 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 160. Υπέρ. Κατά. Εγώ θα έλεγα πως απορρίπτεται. 161. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. 161 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 162 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά γκρίνεται. 163 υπέρ κατά απορρίπτεται 164 υπέρ κατά απορρίπτεται 165 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά κατά Γκρίνεται. 166 υπέρ κατά, κατά. εγκρίνεται 167 υπέρ κατά υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 167. Να το ψηφίζουμε, ναι. Υπέρ, του 167, κατά, απορρίπτεται. 168, υπέρ, υπέρ. κατά, απορρίπτεται. 161, υπέρ. υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά απορρίπτεται 171 υπέρ κατά εγκρίνεται 172 υπέρ κατά απορρίπτεται παράγραφος 48 δεν ψηφίζουμε 173 υπέρ κατά απορρίπτεται. 174 δεν ψηφίζεται, 175 υπέρ. Κατά απορρίπτεται, 176 υπέρ. Κατά. Θα έλεγα πως εγκρίνεται. 177 υπέρ. υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 178 υπέρ. υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στην 184 υπέρ κατά απορρίπτεται. 185 υπέρ κατά απορρίπτεται. 186 υπέρ κατά εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά εγκρίνεται 188 υπέρ κατά εγκρίνεται 189 υπέρ κατά, κατά εγκρίνεται 190 υπέρ κατά εγκρίνεται 191 υπέρ κατά, κατά. απορρίπτεται 192 υπέρ κατά απορρίπτεται 193. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 199 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 200. Είναι απλά, έχει αποσυρθεί. 201 υπέρ Α, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, 201 λοιπόν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 202 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 203 υπέρ. Όχι, όχι, άλλο λάθος. 204. Έχει ε, αποσυρθεί. 204 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 205 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 206 υπέρ. Κατά. Όχι, 207 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 208 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 210 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 211 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 212 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 213 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 214 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 216 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 215 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά ε, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. Τώρα η 221 υπέρ. Α, όχι, έχει αποσυγχωρηθεί. Η καταπίπτει. 224 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 225 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 226 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 227 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 228 υπέρ, Κατά. Εγκρίνεται. 229 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 230 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 231 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 232 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ε, Παύλα 1 υπέρ. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Α. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Α. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη υπέρ 48, 6 κατά 6 αποχές συγχαρητήρια στον εισηγητή. Λιοψηφία. Ταξίζατε τα χειροκροτήματα μετά από τόσο έντονη ψηφοφορία. Ναι, παρακαλώ. Υπάρχουν παρεμβάσεις. Ποιος, τι... Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι εμείς από την ΚΟΕ ε, θέλουμε ψήφ, ε, ψηφο, έκθεση μειοψηφία έχουμε συντάξει, το είπα, τα κατάφερα και θα σας την υποβάλουμε. Από πλευρά της ΓΚΟΕ, μειοψηφούσα άποψη. Για την Ολομέλεια εννοείται προφανώς. Α, θαυμάσαι. Ωραία, σήμερα ψηφίζουμε το εδώ και στην Ολομέλη κάντε ό,τι θέλετε. Θα έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε με την έκθεση για την ΚΕΠΑ. Και έχουμε την τροπολογία 21 υπέρ κατά, κατά απορρίπτεται. Θα σας παρακαλούσα όμως να σηκώνετε τα χεράκια σας γιατί αν δεν βλέπω θα πρέπει να μαντέψω και θα χάνουμε χρόνο με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και άλλα τέτοια. Λοιπόν, 22 υπέρ. Sì, allora, mi viene detto dal segretariato che forse non δεν ξέρετε τι ψηφίζουμε. Λοιπόν, να σας το ξαναπώ. Ψηφίζουμε την έκθεση για την ΚΕΠΑ που σας διαβεβαιώνω εγώ ο Πρόεδρος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εισηγητή, που είμαι εγώ ο ίδιος, εκμεταλλεύομαι και την κατάσταση. Λοιπόν, ψηφίσαμε την πρώτη τροπολογία και στη δεύτερη τροπολογία θα περάσουμε στην τρίτη... Ο κύριος Νταφ. Συγγνώμη. Είμαι ευγνώμων που μας διευκρινίσατε τι ακριβώς κάνουμε. Αλλά μήπως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από την mm. αρχή. Μάλιστα, ξεκινάμε από την τροπολογία 21 ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 29. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροποφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία προφορική 2 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 38 υπέρ, Κατά. Κατά. Σαρανταένα, οι άλλες έχουν ε, καταπέσει, υπέρ, κατά. κατά. Απορρίπτωτε, Συμβαστική. Ηλεκτρονική ψηφοφορία δοκιμαστική για τη για, μάλλον για επιβεβαίωση 41. Για τη 41. Ναι συγγνώμη, συγγνώμη, περιμένετε, περιμένετε. Οκτώ ακόμα δεν έχετε ψηφίσει. Τρει δεν έχετε ψηφίσει. Τρει που μάλλον έχουν πάει για καφέ. Και ένα λιγότερο γιατί έβγαλε την κάρτα. Λοιπόν, τέλος ψηφοφορίας. 28. 29, 28. 28 όχι, 29 ναι. Μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. Στο photo finish βγήκε εδώ. Λοιπόν, η συμβεβαστική 3 υπέρ κατά. κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 44 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 45 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 47 καλύπτεται από την συμβαστική τροπολογία. Οπότε, α, ναι, στις 46, 46, δηλαδή 47 τώρα πάμε, ωραία. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Allora, apriamo la votazione elettronica di controllo. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, ελέγχουμε τη 47. Τροπολογία 47. Quattro persone che non hanno votato. Questo è un argomento che non riesco. Μερικοί δεν ψηφίσαν. 27-28 πέρασε. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49 υπέρ. Κατά. Κατά. Έγκρινεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά, εγκρίνεται. Πάμε στην 50. Υπέρ κατά ε, συγγνώμη, απορρίπτεται. Ο κύριος θέλει να παρέμβει. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας προτείνω κάτι. Ελπίζω να συμφωνεί η Επιτροπή. Η πληροφορική τροπολογία στην παράγραφο 8 ως προσθήκη του θα έλεγε τα εξή. Επαναλαμβάνει ότι η θέση σε ισχύ και η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσία εξωτερική δράση θα πρέπει να γίνουν με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των δημοκρατικών και δημοσιονομικών που αναλογούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. C'è Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Είστε υπέρ. Ωραία. Υπέρ, κατά. Κανείς. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν. Μια δηλαδή, διοθετήθηκε μα και όλες πάμε στη 50. Στην 53 πάμε σε δύο κομμάτια, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, κατά. Δεύτερο τμήμα της 53 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 54 και εδώ δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απο... Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προχωράμε στο 58. Υπέρ. Κατά. Κατά. Απορρίπτεται. Ε, ναι, το περίμενα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 58. Ψηφίζουμε. Α, ένα μόνο che δεν vota, magnifico. Allora Chiudiamo la votazione. 23 a 35 è approvato. Λοιπόν, 35 υπέρ 23 κατά εγκρίνεται. Καλά κάνατε λοιπόν που ζητήσατε επαλήθευση. Πάμε στην παράγραφο 61. Στην τροπολογία 61 δηλαδή. Ε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική έξι. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως έχει γίνει μια μικρή αλλαγή και αντικαθίσταται η φράση υποβαθμίζει την ε, συνοχή και συνέπεια με το αποδυναμώνει την ανεξαρτησία. Αυτή είναι η αλλαγή που έχει γίνει και την οποία υποβάλλω στην δική σας έγκριση. Συμβιβαστική 6 με αυτή τη μικρή αλλαγή που είναι σχεδόν μόνο λεκτική. Λοιπόν, τροπολογία συμβαστική 6 με αυτή την αλλαγή υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην 68, γιατί έχουν καταπέσει οι υπόλοιπες τροπολογίες. Υπέρ. Κατά. Κατά. Απορρίπτεται. 68 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Solito giallo del eh, collega Dormiente. 26 a 32 favorevole. 32 υπέρ, 26 κατά. Οπότε εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, κατά εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά. Εγώ λέω ότι απορρίπτεται.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 Κατά. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 78. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Allora, voto elettronico sul 78. Si apre la votazione. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 78 ψηφίζουμε. passa 78. Περνάει 78. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Κατά. Εγκρίνεται. 79. Υπέρ. Κατά. Κατά. Απορρίπτεται. Α, όχι, συγγνώμη, 80 και, 80, 80 και 81 καταπίπτουν ε, λόγω της συμβαστικής 7. Πάμε στη συμβαστική 8. Η συμβαστική 8 απαιτεί μια σύντομη διευκρίνηση. Ψηφίζουμε σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, όλο το κείμενο χωρίς την έκφραση and Gender Balance. Ψηφίζουμε λοιπόν για το κείμενο χωρίς αυτή την φρασούλα. Υπέρ. Κατά. Κατά. Θα έλεγα πως εγκρίνεται, λοιπόν. Και τώρα θα ψηφίσουμε χωρίς τα το δεύτερο τμήμα, με τη φρασούλα αυτή δηλαδή. Υπέρ. Κατά. Κατά. Εγκρίνεται. Ωραία. Πάμε στην 86. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Questo non l'ho proprio visto, eh. Ε, τώρα δεν μπορώ να δω, λυπούμε, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε. 86 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. είμαστε 61 ψήφισαν, μπράβο όλοι. Απορρίπτεται όμως γιατί ήταν 25 μόνο υπέρ. Λοιπόν, η επόμενη, ε, υπέρ κατά, 88 υπέρ κατά, απορρίπτεται. 89 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτον ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα. Ψήφι πέ. Ψήφι κατά. Εγκρίνεται. Έχουμε την 90 τώρα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 91. Ψήφι πέ. Κατά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εάν δεν σηκώνετε τα χέρια σας, τι να κάνω κι εγώ. Λυπάμαι. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 91, παρακαλώ, της κυρίας Κοπά. Πέρασε. 25 κατά, 35 υπέρ εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 93 επέ. Κατά. Απορρίπτεται 94 επέ. Κατά. Απορρίπτεται 95 επέ, Κατά. Εγκρίνεται. 96 επέ, Κατά. Εγκρίνεται νομίζω. Συμβαστική νέα, Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η συμβαστική, η προφορική συγγνώμη 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι Κατά το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και το δεύτερο και το πρώτο. Ερχόμαστε τώρα στην συμβαστική παριθμό 10. Ψήφι Κατά. Εγκρίνεται. Οι 107, γιατί έχουν καταπέσει οι ενδιάμεσες, ψήφι περ. κατά, εγκρίνεται. 108, ψήφι κατά. Α. Δεν μου σηκώνεται χέρια. Τι να κάνω. Ε, θα την ελέγξω ηλεκτρονικά την 108. Αφού δεν βλέπω τα χέρια σας να σηκώνονται. 108. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. 61 ε, ψήφισαν, 28 υπέρ, 31 ε, κατά, απορρίπτεται. 109 ψήφι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η συμβαστική παριθμών 11, τρία τμήματα. Τμήμα πρώτον, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Το τρίτο, υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. Σε αυτό εδώ το σημείο καταπίπτουν όλες μέχρι την 118 που ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 119. Ναι, ναι. Ναι. Απερίφθη. 119. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 120. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Νο από κάτω, όχι. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 120. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Είναι ένας που έχει βάλει κάρτα αλλά δεν ψηφίζει. Εγκρίνεται 34-26. 121 υπέρ κατά εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά απορρίπτεται. 124 υπέρ κατά απορρίπτεται. 125 δηλαδή 26 διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 127 υπέρ Συγγνώμη, 127 είπαμε. Ναι, έχει καταπέσει η άλλη. 127 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά, καταπίπτει 128 διότι πέρασε 127. Μάλιστα, διορθώνω. Η 128 καταπίπτει διότι εγκρίθηκε 127 η προηγούμενη τροπολογία. Οπότε περνάμε στην 129 που θα ψηφίσουμε σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον, ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Κατά. Απορρίπτεται. Η προφορική υπαριθμό 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 130 είπε. Κατά. Απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Κατά. Εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 134. Έχει αποσυρθεί. 135 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η... Το δεύτερο τώρα τμήμα, πάντα στην 135 είμαστε ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η προφορική υπαριθμών 6 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ορίστε. Λοιπόν, φτάνουμε στη συμβαστική υπαρθμό 12 και εδώ θα ζητήσουμε χωριστή ψηφοφορία. Δηλαδή, θα ψηφίσουμε μέχρι τη λέξη στρατηγική συνεργασίας. Και μετά το υπόλοιπο της παραγράφου. Το πρώτο μέχρι εκεί που σας είπα, μέχρι τη στρατηγική συνεργασία, στην παράγραφο 27. ψήφιπε Κατά. Μα κυρία, ε, μάλλον εγκρίθηκε. Και το δεύτερο, το υπόλοιπο της παραγράφου, ψήφιπε Κατά. Εγκρίνεται. Οπότε και θα περάσουμε στα 138 ψήφι πέρα. Κατά, εγκρίνεται. Η προφορική παριθμόν 7. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε αλλαγή και σας υποβάλλω προς ψήφιση. Προοπτικές ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι τελευταίες λέξεις και αλλάζει και αυτό και γίνεται ευρωπαϊκή προοπτική, αν συμφωνείτε. Αντί για προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό να γίνει ευρωπαϊκή προοπτική. Συμφωνείτε με αυτή τη μικρή αλλαγή. Ωραία, θαυμάσια. Το πρώτο τμήμα έχουμε λοιπόν και ψηφίζουμε την προφορική υπαρθμονευτά. 7, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, με αυτή την αλλαγή που σας είπα, υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. Έχει αποσυρθεί 139, συμβαστική 13 τώρα. Εδώ έχω μια μικρή αλλαγή, τελευταία είναι, ε, τελευταία όμως. Μικρή αλλαγή σας προτείνω. Στην 7η σειρά που λέει «Η αμοιβαίο σεβασμό», «mutual respect», εκεί προσθέτω και την αμοιβαιότητα εγώ, «and πρόσιτη, αν συμφωνείτε, με αυτή τη μικρή αλλαγή. σεβασμό και αμοιβαιότητα. Εντάξει. Το ψηφίζουμε αυτό. Με αυτή τη μικρή αλλαγή, τη συμβαστική 13 ψήφι, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 146. Πάλι σε χωριστά τμήματα. Τμήμα πρώτον, υπέρ. Κατά. Απορρίπτε Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 151. Καταπίπτει. 152 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 153 σε χωριστά τμήματα. Πρώτον υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα είπε. Κατά. Απορρίπτεται. 154 είπε. Κατά. Απορρίπτεται. 155. κατά, πίπτη και έχουμε. Την 156 ψηφιπέ, Κατά. Θα με συμπαθάτε, αλλά δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε την 156 ηλεκτρονικά, σας παρακαλώ. Αν δεν σηκώνετε χέρια, δυστυχώς θα πρέπει να ζητάω ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έτσι, εμβάθυνση κάπως, αν δεν έχουμε άρση των χείρων. Δύο μου λείπουνε. Δεν ξυπνάνε, τι να κάνω μάλλον 31 υπέρ 26 κατά, ε, εγκρίνεται. 157 πίπτη, 158 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η προφορική υπαριθμών 8 τώρα, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 160 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 165. Δεν την ψηφίζουμε διότι εγκρίναμε την προηγούμενη. 166 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 167 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτον. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Θα έλεγα εγώ. Α, καλά δεν λέω. Τότε να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Ε, της 167 αρχίζει το ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όλο μας λείπει ένας παρόν κατά τα άλλα όμως. 38-24 ε, εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά. Τι έγινε με την 179. Α, ζητώ συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Δεν ψηφίζουμε την 168 διότι είναι ταυτόσημη με την 179. Πάμε στην 169. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η προφορική τώρα υπαριθμών 9 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 170. Δεν ψηφίζουμε ούτε την 171 και πάμε στην 173. Ψηφί υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 178 κατά πίπτη. 180 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 181 υπέρ. Ε. Κατά. Απο... Ε, εγκρίνεται, συγγνώμη. Και τώρα πάμε σε αιτιολογικές σκέψεις. Η... Τρία υπέρ. Ε. Κατά. Αποχές. Σε δύο τμήματα ή τέσσερα τώρα. Το διατηρητική σκέψη α. Υπέρ του πρώτου τμήματο. Κατά. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η πέντε υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 18 λέει ο Πρόεδρος, αλλά είναι 14. Ε, ζητώ συγγνώμη, 14. Ε, ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνεται και περνάμε στην 7 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Τροπολογία παριθμών 7 στο Β. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 9. Ε, καλύπτεται. Πάμε στη 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 10, προφορική. Ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Κατά. Εγκρίνεται. Ναι. Και τώρα θα πάμε στη 13. Ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Είμαστε στην εντυπωσιακή σκέψη Δέλτα. Κατά. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 16. 16 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αφήνουμε το 20 λοιπόν που έχει καλυφθεί και πάμε στην 1 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την ψηφοφορία σχετικά με τον προϋπολογισμό, δηλαδή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμού, για να το πω ακριβέστερα. Τροπολογία 1 υπέρ. Να τις κάνουμε όλες, ναι, όχι χωριστά είναι χωριστά, θα τις, τις ψηφίσουμε. Λοιπόν, budget 1 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Προϋπολογισμού 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προϋπολογισμού 8 υπέρ. Κατά. Εποχές. Ε, εγκρίνεται. Προϋπολογισμού 9 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Προϋπολογισμού 10 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τελική και ολοκληρωτική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. πάλι τρει δεν ψήφισαν ενώ έχουν βάλει κάρτα. Τι να κάνω. Λοιπόν, 51 υπέρ, 4 κατά μία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, ε, ένα τον ίδιο δηλαδή. Μάλιστα, μάλιστα. Ο κύριος Βίλι Μάγερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως είχα την ευκαιρία να εκδηλώσω στη συνεδρίαση των συντονιστών, σας λέω ότι η ομάδα μου θα καταθέσει έκθεση μειοψηφία, γιατί απέχουμε πόρο από τη φιλοσοφία της έκθεσης που μόλις εγκρίθηκε στην Επιτροπή μας. Συγχαρητήρια σε εσά προσωπικά, αλλά δυστυχώς αυτή τη φορά ατυχήσαμε. Συνήθως σας συγχαίρω, αλλά τώρα σας ευχαριστώ. Καλοσύνη σας. Σέβομαι τη σκέψη σας, έχουμε εδώ την άλλη άποψη της πλειοψηφίας, αλλά βεβαίως και μπορείτε να φέρετε στην Ολομέλεια έκθεση μειοψηφίας, όπως ακούστηκε και προηγουμένως και το έχετε δηλώσει. έχουμε... την έκθεση Γκάλερ για την απαλλαγή. Μία μόνο τροπολογία υπάρχει για την απαλλαγή 2008 2008-2003. Υπέρ της μοναδικής τροπολογίας, κατά εγκρίνεται. Ηλεκτρονική συνολική ψηφοφορία. Πάλι μερικοί. ψήφισαν 54 επί 57 παρόντων, τέλος πάντων. 53 ψήφισαν. 50 υπέρ, 3 αποχές, μία ψήφος κατά. Λίγουν οι σημερινές ψηφοφορίες. Τώρα έχουμε το Προεδρείο που θα αρχίσει αμέσως σε λίγο. Μόλις αδειάσει η αίθουσα από όσους